Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε αυτή την κοινή συνδιάσκεψη για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας καλωσορίσω σήμερα σε αυτή την αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. είναι εδώ και η κυρία Τόνι Σμιτ. Να σας καλωσορίσω και εσάς, κυρία Πρωθυπουργέ της Δανίας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπαρόζο. Κάθεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα. Αυτό αποδεικνύει τη στενή συνεργασία που έχουν τα τρία θεσμικά όργανα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι πρόεδροι τους. Είναι, έχουμε μια πραγματική πρόθεση για πάρα πολύ στενή συνεργασία. Η Ευρώπη, αγαπητοί, αγαπητές και κύριοι, βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση. Βρισκόμαστε σε μια κρίση χρέους. Παντού υπάρχουν περικοπές. Όλο και περισσότερη οικονομία πρέπει να γίνει. Αλλά κάτι είναι ξεκάθαρο. Δεν θα γίνει αποδεκτό ένα μικρότερο ποσό για το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό ενδεχομένως για κάποιους ακούγεται παράλογο ή ανεύθυνο, αλλά είναι κάτι... Αλλά ισχύει το αντίθετο. Είναι και υπεύθυνο και λογικό. Ε, ήταν εύκολο να καταλάβουμε ότι ήταν ευρωβουλευτέ αυτοί που μόλι χειροκρότησαν. Και ακούω ότι χειροκρότησε και ο Υπουργό Οικονομικών από το Βραδεμβούργο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να ζητά κάποιος περίπλο. Ε, περικοπές στο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά δεν είναι κάτι λογικό. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θέλουν να εξοικονομήσουμε στο, κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί στην περισσότερη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ιδίω τώρα, εφόσον το 2013 λύγει το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να την το επόμενο, το Κοινοβούλιο βαίνει καλώ προετοιμασμένο σε αυτέ τι ε, προετοιμασίε. Ήδη τον Ιούνιο του 2010 δημιουργήσαμε μια ειδική επιτροπή ένα χρόνο πριν η Επιτροπή να, να κάνει την πρώτη της ε, πρόταση. 8 Ιουνίου 2011 αυτή η Ειδική Επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε την έκθεσή του για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η έκθεση έχει να κάνει με τις πολιτικές μας προτεραιότητες και προτείνει μια δομή για, την ε, μεσοπρόθεσμη, για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό λέει πόσα χρήματα χρειάζεται, απαιτεί να επιστρέψουμε στο σύστημα των ιδίων πόρων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας όρος που πολλές φορές δεν είναι γνωστός ούτε στους Υπουργούς Οικονομικών, παραδόξως. Και να επιστρέψουμε λοιπόν στους ίδιους πόρους χωρίς ειδικέ ρυθμίσεις γιατί λοιπόν αρνούμαστε ιδιαίτερα σε αυτά τα πλαίσια της κρίσης αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη μόνο με έναν σωστό προϋπολογισμό μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γιατί η Ευρώπη μόνο με έναν σωστό προϋπολογισμό μπορεί όλα τα σημαντικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί να τα αντιμετωπίσει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε τις προκλήσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και την απασχόληση να τις αντιμετωπίσουμε με έναν σωστό προϋπολογισμό. Το να παγώσουμε τον προϋπολογισμό ή να τον περικόψουμε δεν βοηθάει κανέναν για να βγει από την κρίση. Χρειαζόμαστε τις επενδύσεις στις περιφέρειές μας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των ανθρώπων μας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στους ανθρώπους της περιφέρειας και της περιφέρειας για να κινητοποιήσουμε την οικονομία μας. Δεν λειτουργεί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνέχεια σε όλες τις συναντήσεις τους να καθορίζουν επιπρόσθετα καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα κάθε φορά να περικόπτουν το ποσό για αυτά τα καθήκοντα. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε τις φιλόδοξες ε, πολιτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέμε να φτιάξουμε μαζί και έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να είναι μια προστιθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Γιατί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επενδύουμε στους τομείς όπου υπάρχουν στα κράτη-μέλη περικοπές. Το συμφέρον των πολιτών είναι κάτι που θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη στις επόμενες διαπραγματεύσεις και θα το υπερασπιστούμε με δύναμη. Οι εκπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν κατά τη διάρκεια της ε, προετοιμασίας της, ε, της, ε, του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου να λειτουργούν επίσης όρις με τους συναδέλφους από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου και κυρία Πρωθυπουργός ανήκει σε αυτούς, γιατί ξεκίνησαν ανεξάρτητα αυτές τις εργασίες και συμφώνησαν πάρα πολύ νωρίς. Και ήταν ένα πάρα πολύ θετικό σήμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε μια εντολή διαπραγμάτευσης. Έχουμε την έκθεση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε μια ομάδα διαπραγμάτευσης με έμπειρους εμπειρογνώμονες επί θέματα προϋπολογισμού. Έχουμε μια ομάδα επαφής μέσα στο Κοινοβούλιο για να υπάρξει και μια σωστή δομή εσωτερικής επικοινωνίας. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει και ένα θεσμικό ρόλο όπου συναντιέται με τους πρόεδρους του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής, επίσης όρης. Σήμερα είναι μια τέτοια συνάντηση, όπου και τα τρία θεσμικά όργανα προσπαθούν να συμφωνήσουν με, για τις θέσεις τους. Θα ήθελα να πω στους δύο συναδέλφους μου εδώ πάνω ότι αυτό το καθήκον το παίρνω πολύ στα σοβαρά. Για μένα δεν είναι απλώς κάτι τυπικό, αλλά είναι ένα από τα αποφασιστικά καθήκοντά μου ως πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι με πάθος αφιερώνομαι στα καθήκοντά μου. Και να είστε έτοιμοι, αυτό θα κάνω και τώρα. Οι εκπρόσωποι των πολιτών έχουμε δικαίωμα ψήφου και αυτό το δικαίωμα θα το εκμεταλλευτούμε. Το περιεχόμενο της πολιτικής, ωστόσο, είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί από τους εμπειρογνώμονες. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν, δεν συμμετέχει σε διαδικασία συνένεσης, αλλά συναπόφασης. Και λέω ξεκάθαρα ότι αυτό το δικαίωμα της συναπόφασης θα το υπερασπιστούμε. Όλες οι προσπαθ, προσπάθειες, ζητήματα πολιτικής, ε, να τα να αφήσουμε να τα αποφασίσουν αμέσως οι Υπουργοί Οικονομικών και μετά να, να μην υπάρξει το δικαίωμα της συναπόφασης του Κοινοβουλίου είναι κάτι που εμείς δεν θα το δεχτούμε. Αυτό δυστυχώς πρέπει να το πω ευθύ εξ αρχής. Και ελπίζω να, τώρα που το είπα να είναι και ξεκάθαρο. Να σας πω και κάποια πράγματα για το σημερινό πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, Χρειαζόμαστε έργασης και ανάπτυξη για να βγούμε από την κρίση. Όταν δώσουμε στον άνθρωπο ένα σίγουρο μέλλον, χρειαζόμαστε, για να του δώσουμε αυτό το μέλλον χρειαζόμαστε επενδύσεις. Τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία των πολίτη θα, θα την βρούμε όταν υπάρχει ένα σωστός ευρωπαϊκός και εθνικός περιπολογισμός. Όταν λοιπόν τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται ακριβώς στα σημεία όπου τα κράτη-μέλη είναι αναγκασμένα να κάνουν περικοπές. Για το πού θα επενδύσουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο τρόπο, αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα. Ωστόσο, δεν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, θέλουμε το αντίθετο, από κάτω προς τα πάνω. Και γι' αυτό αυτή τη λειτουργία επιτελεί και αυτή η συνδιάσκεψη εδώ με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν θέλουμε να κρατιόμαστε δογματικά σε κάποιους προκαθορισμένους αριθμούς, αλλά θέλουμε μια καλώς προσανατολισμένη συζήτηση. Υπάρχουν κράτη που θέλουν να εξοικονομήσουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ και παρόμοια ποσά. Αλλά ενδεχομένως να μην μπορέσουν και τα υπόλοιπα κράτη να αποφύγουν το να υπάρξει λιγότερη ανάπτυξη περιφέρειας, να υπάρξουν λιγότεροι φοιτητέ στο Εράσμος. Οι τομείς επιτυχίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι τομείς που πλήττονται περισσότερο από αυτό το εγχείρημα. Και αυτό ενδεχομένως θα σας εκπλήσει αν εμείς στο Κοινοβούλιο λέμε ότι εμείς τέτοιου είδους πολιτική δεν θέλουμε να την υποστηρίξουμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε επίσης ότι το, ο προϋπολογισμός της Ένωσης μεγάλωσε πολύ λιγότερο από ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί στα κράτη-μέλη. Αυτός είναι ένας αριθμός που σας παρακαλώ να το ξανασυζητήσετε, το πόσο αυξάνονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί που αυξάνονται πολύ περισσότερο από ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Και γι' αυτό το λόγο πολλές κατηγορίες ενάντια στον ευρωπαϊκό πολιτισμό δεν ευσταθούν. Τώρα κάτι για τους ίδιους πόρους. Η έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο λέει ότι υπάρχει μια στενή σχέση εδώ ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα και γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε και για τους νέους ίδιους πόρους εδώ. Ένα πραγματικό σύστημα ίδιων πόρων προβλέπεται στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. μετά το άρθρο 311 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, το 311 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι η παράγραφος 11 του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά η Συνθήκη της Ένωσης. Το ότι, αυτή, το ότι αυτό το άρθρο είναι τόσο άγνωστο, θα ήθελα, επειδή είναι τόσο άγνωστο, θα ήθελα να σας το διαβάσω αυτό το άρθρο. Η Ένωση εξοπλίζεται με τα απαραίτητα μέσα για να πετύχει τους στόχους της και να μπορέσει να υλοποιήσει την πολιτική της. Ο προϋπολογισμός, άσχετα από τις λοιπές, ε, από τα λοιπά έσοδα, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Αυτό είναι το άρθρο 311 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα μέλη, από ό,τι ξέρω. η εφαρμογή, η χρήση των ιδιών πόρων θα σταματήσει αυτή την πολεμική. Και γι' αυτό χαιρετίζω τις νέες προτάσεις της Ένωσης. Χαιρετίζουμε τις ε, νέες προτάσεις της, ε, της Επιτροπής ε, για, την, για, για τον φόρο των θρηματοπιστωτικών συναλλογών και του ΦΠΑ. Το να μην υπάρξει συζήτηση επί αυτών των θεμάτων δεν είναι ένας τρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρέπει να τα συζητήσουμε όλα Τώρα, αν θα συζητήσουμε, το, το, θα, θα συμφωνήσουμε στο τέλος είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Όλα αυτά τα σημεία βρίσκονται στην ημερήσια μας διάταξη. Και εσείς κυρίες και κύριοι ως εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Εθνικών Κυβερνήσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά αυτά τα ζητήματα σήμερα το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευθύνη προσεγγίζει αυτή τη συζήτηση. Και στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα, την καινοτομία. Και βλέπουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε ένα εργαλείο για την διασφάλιση του μέλλοντος των Ευρωπαίων πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επίτροπης μου είπε πριν από αυτή τη συνάντηση να είσαι σκληρός αλλά φιλικός. Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στις προσδοκίε. του. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρωθυπουργός. Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Σούλτ, πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Μπαρόζο, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, υπουργοί και επίτροποι, κυρίε και κύριοι. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα, εξ ονόματο τη Δανική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να επεκτείνω τι ευχαριστίε μου προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί τη σημερινή εκδήλωση. Επίση, ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη στενή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και όλα αυτά οδήγησαν βεβαίω και στη σημερινή συνδιάσκεψη. Επίση, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω τόσου πολλού εκπροσώπου από τα Εθνικά Κοινοβούλια γνωρίζω από την προσωπική μου εμπειρία το πόσο σημαντική είναι η στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια σε όλους τους τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, ως πρόεδρος Συμβουλίου σας ε, διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να συνεργαστούμε στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σήμερα εδώ έτσι ώστε να σημειώσουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι οι διαπραγματεύσεις ε, λαμβάνουν χώρα σε μια χρονική στιγμή όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια πήραμε σημαντικές ε, αποφάσεις ε, ε, και κρίσιμες αποφάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο με στόχο να αντιμετωπίσουμε την κρίση του δημόσιου χρέους. Σημειώσω μεγάλη πρόοδο, αλλά τα δημόσια νομικά των κρατών μελών εξακολουθούν να υφίστανται πίεση και η δημοσιονομική εξυγίανση θα εξακολουθήσει να είναι μια σημαντική πρόκληση στα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν χρειάζονται πολλά χρόνια για να χάσει κανείς την οικονομική του αξιοπιστία, αλλά χρειάζονται δεκαετίες για να την επαναπακτήσει. Ταυτόχρονα παρατηρούμε βραδία ανάπτυξη και αύξηση της ανεργίας, κυρίως της ανεργίας των νέων. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμό από τις αναδυόμενε οικονομίες και το δημογραφικό πρόβλημα ε, είναι δύο άλλες προκλήσεις ε, που έρχονται να προσθεθούν σε αυτές που ήδη αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό είναι ύψη τη σημασία να επιταχύνουμε την ε, ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Επίση είναι σαφέ ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις ούτε θαυματουργές λύσεις. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι το επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα μας δώσει ε, μια χρυσή ευκαιρία για να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε τον προπολογισμό έτσι ώστε να είναι ε, καλύτερα ευθυγραμμισμένος με τις ε, μελλοντικές ανάγκες και ότι πραγματικά θα υπάρξει αλλαγή και στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρώπη. Κάθε 7 χρόνια μα δίνεται ευκαιρία να ε, αλλάξουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε λάθο. Οι διαπραγματεύσει για το, πολιτεύσιο για, το για το δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον προπολογισμό αποτελούν μια ευκαιρία για μα ε, ω πολιτικού για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, προσφέρει λύσει στα δύσκολα προβλήματα ε, παρά την οικονομική κρίση που διανύουμε. Δεν έχω καμία αυταπάτη και πιστεύω και εγώ ότι οι διαπραγματεύσει θα είναι δύσκολε. Το διακύβευμα είναι υψηλό. Και όλοι το γνωρίζουμε. Και ε, εδώ ε, στη συζήτηση υπησέρχονται τεράστια χρηματικά ποσά. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι πλευρές κάθονται στο τραπέζι με τα δικά τους επιμέρους συμφέροντα. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όμω σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να επιδείξουμε όλη την πολιτική βούληση και το θάρρος έτσι ώστε να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος. Θέλω να είμαι σαφή. Η τελική συμφωνία για το, δημοσι... το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι ε, κάτι το εύκολο. Αυτό ήταν ξεκάθαρο για αρκετό καιρό. Ήταν ξεκάθαρο, δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία επί προεδρίας. Προεδρία. Σα διαβεβαιώνω όμω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδο στι διαπραγματεύσει κατά τη διάρκεια τη δική μα Προεδρία. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχο μα είναι να αναπτύξουμε μία βάση, να υπάρξει μία βάση για το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να συζητηθεί η βάση αυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2012. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε θα χαράξουμε τον δρόμο έτσι ώστε να υπάρξει τελική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Η Δανική Προεδρία εργάζεται σκληρά στα πλαίσια της εντολής που εδόθη στη Δανία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2011. Για την εκπλήρωση τη εντολή αυτή, ήδη έχουμε ξεκινήσει τι προκαταρκτικέ συζητήσει σε επίπεδο υπουργών. Ο στόχο μα είναι να μειώσουμε το κενό και τι διαφορέ ανάμεσα στι θέσει των αντιπροσωπιών έτσι ώστε ε, να υπάρξει ε, βαθμιαία ε, συμφιλίωση των διαφορών. Αυτό είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και να υπάρξει μια συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012 ε, κατά μείζον λόγο, διότι η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί απαραίτητη προπόθεση έτσι ώστε να περάσουμε στι επίσημε διοργανικέ διαπραγματεύσει που θα ολοκληρώσουν το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τώρα όμω η Δανική Προεδρία ε, έχει ξεκινήσει στενέ και τακτικέ επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα επίπεδα και θα ξεκολουθήσουμε να το πράττουμε. Ο στενό διάλογο ανάμεσα στα όργανα καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία αυτή είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να υπάρξει συμφωνία. Πιστεύω πιστεύω ότι η σημερινή συνδιάσκεψη σήμερα, η συνδιάσκεψη αυτή υψηλού επίπεδου, συμπληρώνει τον συνεχιζόμενο διάλογο που αποτελεί το στόχο μα, διότι με τον τρόπο αυτό οι βασικοί εμπλεκόμενοι στι διαπραγματεύσει έχουν μία ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψει με ανοιχτό και επικοδομητικό τρόπο. Ακριβώ γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα. Και όπω σα είπα και προηγουμένω, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου ε, προ τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, προ όλου εσά που ήρθατε σήμερα εδώ πιστεύω ακράδαντα ότι η δική σας συμβολή που στηρίζεται σε πλήρη γνώση της ε, οικονομίας ε, των κρατών μελών και της πολιτικής πραγματικότητας ε, στη χώρα σας. Η συμβολή σας λοιπόν στη σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να μας κάνει όλους να καταλάβουμε τις, τις θέσεις όλων μας και να χαράξει το δρόμο για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα όργανα που θα λάβουν χώρα στο δεύτερο ήμιση του 2012. Το βασικό ζήτημα της σημερινής συζήτησης είναι φυσικά το εξής πώς θα πρέπει να είναι στο μέλλον ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλές απόψεις ε, σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας ε, ε, μεταφέρω ορισμένες απόψεις για τις αρχές που κατά την άποψή μου θα πρέπει να καθοδηγούν την περαιτέρω εργασία μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση υποστηρίζει την ατζέντα για την ανάπτυξη δημιουργία θέσεων εργασία με καλύτερο τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα. Αυτό απαιτεί πολιτικό θάρρο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε συνεχίσουμε τα κονδύλια στι πολιτικέ που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα τη Ευρώπη αλλά και την ανταγωνιστικότητά τη. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι η ενίσχυση ε, των προσπαθειών μα στον τομέα ε, έρευνα και καινοτομία, διαμέσου του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμη ε, σημασία για την ανταγωνιστικότητά μα στην παγκόσμια οικονομία. Δεύτερο, χρειαζόμαστε ένα πιο πράσινο προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πράγματι, η σημασία τη κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντο πρέπει να εκφράζεται καλύτερα σε όλα ε, τα σχετικά προγράμματα. Αυτό βεβαίω θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να υποστηρίζει ε, και την ατζέντα για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση που ανέφερα πριν από λίγο. Τρίτον, η αλληλεγγύη θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εστιάσουμε ε, του σχετικού πόρου στην ανάπτυξη των λιγότερο ευημερούντων κρατών μελών και περιοχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, σε αυτή τη χρονική στιγμή όπου ε, σπανίζουν οι πόροι, θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για να δούμε το πώς ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσφέρει πραγματική προσθέμενη αξία και μέγιστο αποτέλεσμα για κάθε ευρώ που δαπανούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια νοοτροπία αποδοτικότητας και αξιολόγηση, όπου η συγκριτική αξιολόγηση και οι δείκτες θα αποτελούν ένα ε, σημαντικό τμήμα των εργαλείων σε όλα τα ε, προγράμματα δαπανών. Και πρέπει να έχουμε το θάρρο να κλείσουμε ή να υποβαθμίσουμε τα προγράμματα τα οποία δεν οδηγούν σε αυτά αποτελέσματα. Επίση, θα πρέπει να επιταχύνουμε τι προσπάθειέ μα για να εξασφαλίσουμε υγιή και πιο αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Πρέπει να δείξουμε στου πολίτε μα ότι τα χρήματα τα οποία δαπανώνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήματα τα οποία δαπανώνται με τον σωστό τρόπο. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να απλοποιήσουμε του κανόνε. Η γραφειοκρατία δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την εξασφάλιση αποτελεσματικών πολιτικών που ε, αποδίδουν όσο το δυνατόν περισσότερο ε, σε κάθε ευρώ το οποίο δαπανάμε. Τέλο, η χρηματοδότηση του μελλοντικού προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διακρίνεται από διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να είμαι ξεκάθαρη. Η δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, δεν σημαίνει μόνο ένα σκεπτικό ε, ε, ίσης ανταπόδοσης, όπου, όπου κάθε κράτος μέλος ε, διακρίνεται από μία έμονη ιδέα όσον αφορά τη δική του καθαρή θέση. Η δικαιοσύνη για μένα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη με ε, ίσα επίπεδα πλούτου σε γενικές γραμμές πληρώνουν τα ίδια ποσά στον προπολογισμό. Η αλληλεγγύη είναι μια σημαντική αρχή ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αυτό τι σημαίνει, ότι οι πιο πλούσιε χώρε θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στον προπολογισμό από ότι οι λιγότερο ευημερούσε. Σε τελευταία ανάλυση, αυτή η αρχή ε, θα ε, είναι προ όφελο όλων μα. Πιστεύω ότι οι αρχές αυτές αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία θα εξασφαλίσουν ένα μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίο θα χαρακτηρίζεται από τι δικέ μα προσπάθειε να επιλύσουμε και να ξεπεράσουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Βεβαίω, αυτέ είναι οι δικέ μου απόψει. Και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η Δανική Προεδρία στην ε, ε, μεταγενέστερη εργασία θα λάβει υπόψη όλε τι απόψει, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα προπολογισμό τη Ευρώπη που να είναι προ όφελο όλων μα. Η σημερινή συνδιάσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία για, για εσά, για του εμπλεκόμενου, για όλου μα, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε αυτέ τι συζητήσει για το ποιε είναι οι πιο σημαντικές αρχές που θα πρέπει να καθοδηγούν το μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί λοιπόν μια σημαντική ευκαιρία για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλοι τι απόψει όλων. Και πραγματικά ελπίζω με όλη μου την καρδιά οι σημερινέ συζητήσει για του νέου ίδιου πόρου και για τι δαπάνε στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα οδηγήσουν σε πιο συγκεκριμένε συζητήσει και σε συγκεκριμένε προτάσει για το πώ θα εξασφαλίσουμε ένα προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μα βοηθήσει να προετοιμάσουμε την Ευρώπη του μέλλοντο. Όπω ήδη σα είπα, εμεί, ω Προεδρία θα ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τη σημερινή συζήτηση. Αποτελούν ε, και θα αποτελέσουν κρίσιμη συμβολή στη συνεχιζόμενη εργασία τη Προεδρία, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα με την προσοχή, για την προσοχή σα και ελπίζω ε, να είναι σημαντικά τα αποτελέσματα τη σημερινή ε, συνδιάσκεψη. Ευχαριστώ. Κύριο Πρόεδρο Μπαρόζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε ε, Σούλτ, κυρία Θόρν Σμίτ, κύριοι Υπουργοί, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητοί κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα καλωσορίσω εδώ εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σούλτ και την Πρωθυπουργό Θόρνινγκ Σμιτ για την εξαίρετη συνεργασία μα για να ε, διοργανώσουμε από κοινού αυτή τη δεύτερη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πολύ ωραίο το γεγονό ότι βλέπω εδώ τόσου πολλού αξιότιμου συμμετέχοντε εδώ. Μεταξύ άλλων εκπροσώπου από το Ευρωκοινοβούλιο και των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και και εκπροσώπους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Εσείς όλοι είστε ε, οι πιο σημαντικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τους ε, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσετε την επιτυχία όχι μόνο αυτής της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, αλλά και το πιο σημαντικό είναι κατά την εφαρμογή των στόχων του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει επένδυση στην ανάπτυξη των οικονομιών μας σε θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. Τελευταίες εβδομάδες υπάρχει λιγότερη πίεση στην ευρωπαϊκή οικονομία και κάποια σημάδια μεγαλύτερη σταθερότητα από ότι ε, το δεύτερο ε, εξάμεινο πέρυσι. Όμως δεν έχουμε εξέλθει από την κρίση και δεν μπορούμε να ε, εφησυχαζόμαστε. με, αυτή την με αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία να δούμε λιγάκι τι ακριβώς χρειάζεται η Ευρώπη. Απασχόληση βιώσιμη απασχόληση. Αυτό που λέμε απασχόληση ευφυή για όλους. Οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να προωθήσουμε αυτή την ανάπτυξη. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι για την ανάπτυξη έχουμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα του 2020. Για τις επενδύσεις έχουμε το Ευρωπαϊκό Πολιετές Πλαίσιο. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί για την Ευρώπη 2020. Είναι μια συνολική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσφάτως επιβεβαίωσε και πάλι τους πέντε στόχους για την Ευρώπη 2020 και επιβεβαίωσε και τις κύριες προτεραιότητες ε, όπως προτείνονται και στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις. Δεν μπορεί να μιλάμε συνέχεια για την ανάπτυξη και να μην είμαστε συνεπείς και να μην προτείνουμε συγκεκριμένα εργαλεία για τις επενδύσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα είναι αποφασιστικέ για την επίτευξη του κοινού μα στόχου, για την δημιουργία μιας οικονομίας ε, ε, συνολικής, που θα του περιλαμβάνει όλους μέσα στα επόμενα χρόνια. Εμείς ε, έχουμε ένα φιλόδοξο εδώ πλαίσιο. Τη στιγμή μάλιστα που οι εθνικοί προπολογισμοί υπόκεινται σε πίεση, αυτό το σχέδιό μας δεν θα κοστίσει τίποτα παραπάνω στους φορολογούμενους. Ταυτόχρονα με τα ίδια κονδύλια θα διασφαλίσουμε ότι θα στοχεύσουμε σε τομείς όπου θα έχει προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή δράση και συμπληρωματικότητα, επενδύοντας στην έρευνα, ε, στα δίκτυα και στην υποδομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δρομολογεί ε, πόρους για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς, για την πρόθεση της αποτελεσματικότητάς μας, αλλά και για τη στήριξη της βιωσιμότητας της οικονομίας μας. Ε, ένα ευρώ που δαπανάται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διάφορα ευρώ συνήθω από του εθνικού προπολογισμού μέσω συνεργειών και αποτελεσμάτων κλίμακα και ε, μπορεί να μοχλεύσει και ιδιωτικέ δαπάνε για να έχουμε μεγαλύτερο συνολικό αποτέλεσμα. Και αυτό διότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι ο προπολογισμό για τι επενδύσει. Επιμένω σε αυτό γιατί ξέρουμε ότι κάπου ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, προβάλλεται ως ο προϋπολογισμός ε, που ε, προκαλεί δαπάνες. Όχι. Εδώ δεν μιλάμε για δαπάνες ή για επενδύσεις για την Ευρώπη, για τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτές οι επενδύσεις επιστρέφουν στα κράτη-μέλη, στους πολίτες μας, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός ο προϋπολογισμός υποστηρίζει σχέδια, έργα και προτεραιότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την στρατηγική περί Ευρώπη 2020. Αυτό το ξέρουμε ότι συμβαίνει και στην πολιτική συνοχή. Και εδώ θα έχουμε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο και απλουστευμένα προγράμματα για να αξιοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές που είναι πολύ σημαντικές σημαντικέ για τι επενδύσεις την απασχόληση και την ανάπτυξη. Όμω, σήμερα θα ε, δώσουμε κάποια βασικά παραδείγματα ε, για τους τομεί που μα ενδιαφέρουν. Έρευνα και καινοτομία, ε, παιδεία και ο μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη. Εκεί θα έχει προσθεμένη αξία ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρώτα απ' όλα, έρευνα και ανάπτυξη η ε, έρευνα αφορά το μέλλον της οικονομίας μας. Έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, με τη δημιουργία των μελλοντικών θέσεων απασχόλησης. Ξέρουμε ότι εκείνες οι χώρες που συνειδητά ε, ε, επένδυαν περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, ε, άντεξαν καλύτερα την κρίση από εκείνε που έμειναν πίσω. Η έρευνα και η καινοτομία δίνει στι εταιρείε μα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ε, γενικότερα αποδίδουν περισσότερο οι θέσει απασχόληση εκεί όπου γίνεται έρευνα, εκεί όπου υπάρχει καινοτομία. Η Ευρώπη θέλει να είναι ο leader σε αυτού του τομεί. Χρειαζόμαστε και ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ε, χωρίς την ευρωπαϊκή κλίμακα, χωρίς την συνέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και ε, στο ίδιο επίπεδο με τους μεγάλους ε, ανταγωνιστές μας στον κόσμο. Τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία και είναι πολύ σημαντικό να ε, χρησιμοποιήσουμε από κοινού τους πόρους μας. Αυτό σημαίνει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες προκλήσεις. Ε, θα, βελτιώσουμε την υγειονομική περίθαλψη, θα ε, προωθήσουμε πιο ε, πράσινες μεταφορές και θα βελτιώσουμε την ασφάλεια και στον τομέα των τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε για να είμαστε πιο καινοτόμοι στην Ευρώπη και ε, να κάνουμε αυτό το άλμα, αν θέλετε, από την ιδέα στην αγορά. Δεν αρκεί να έχει κανεί μεγάλε ιδέε. Θα πρέπει να δημιουργήσει και τι κατάλληλε συνθήκε ώστε όλα αυτά να γίνουν πράξη σε επιχειρήσει, σε θέσει απασχόληση. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξία για την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη. Έχουμε την ε, πρόταση ε, των 80 δι ευρώ που ονομάζεται Ορίζοντα 2020. Πολύ σημαντικό βήμα για το μέλλον. Και περνάω τώρα στην παιδεία. Μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι 35% όλων των θέσεων απασχόληση θα απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση και περισσότερα προσόντα. Ε, θα πρέπει τα εκπαιδευτικά μα συστήματα να να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Εμείς προτείνουμε στη νέα περίοδο το νέο πρόγραμμα «Ο Έρασμος για όλους». Βασιζόμενοι στην επιτυχία και την φήμη του προγράμματος Εράσμους, θα δώσουμε την ευκαιρία σε 5 εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό. Α, διευρύνουμε λοιπόν το πεδίο του Έρασμου και αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν ε, τρέφει την φιλοδοξία να εκπαιδευτουν στο εξωτερικο α διευρυνουμε λοιπον το πεδιο του ερασμου και αυτο σημαινει οτι η κομισιον τρεφει την φιλοδοξια να επενδυσει ε, στα προσόντα ε, και στις ε, δεξιότητες για τους νέους 19 δις προτείνουμε το ώστε να, να υποφεληθεί ο διπλάσιος αριθμός των νέων μας από αυτό το νέο πρόγραμμα. Τα συστήματα εκπαίδευσης είναι και θα παραμείνουν εθνική αρμοδιότητα. Όμως, ε, το να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να εργαστούν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό για να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες, να ανοίξουν νέες πόρτες ε, και να ε, προωθηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η προσαρμοστικότητα η ελεύθερη κυκλοφορία ε, και οι μεταφορές ε, είναι, ε, κρύβονται πίσω από το μηχανισμό Connecting Europe, για τον οποίο προτείνουμε 50 δις ευρώ. Ε, τα εμπόδια δεν μας ε, βοηθούν τώρα να αξιοποιήσουμε πλήρως την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα και να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες ε, να ταξιδεύουν περισσότερο. αυτό θα βοηθήσει πολύ και τις μικρομεσαίες. Ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε τα όρια της παραδοσιακής λογικής, αν θέλετε, των εθνικών προϋπολογισμών και να δημιουργήσουμε μια δυναμική επενδύσεων από την οποία θα υποφεληθεί ολόκληρη η ενιαία αγορά. Ε, οι διασυνδέσεις στον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε ε, ό,τι κάνει το ένα κράτος μέλος να βοηθάει και τις υπόλοιπες. Να δημιουργήσουμε ένα γενικό δίκτυο για τις ανανεώσιμες, για παράδειγμα δεν μπορούμε να προωθήσουμε ε, αυτά τα θέματα αν δεν έχουμε και τα βασικά δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρότασή μας είναι ένα 38 ε, παράδειγμα ε, μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ε, προσέγγισης για να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο μηχανισμός Connecting Europe είναι πολύ σημαντικός. Εκεί τα καινοτόμα μέτρα, τα καινοτόμα εργαλεία θα ε, κάνουν τη διαφορά προσελκύοντας και ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και ε, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο ε, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στις αρχές του μήνα οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρότασή μου για ένα πιλωτικό ομόλογο έργων. Έτσι η Κομισιόν ελπίζει ότι θα προλιάνουμε το έδαφος για πιο συστηματική χρήση ε, αυτού του μέσου μέσω του μηχανισμού Connecting Europe. Ε, τα ομόλογα έργων θα βοηθήσουν για να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα ε, μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης προκειμένου να προωθήσουμε έργα ευρείας κλίμακας και να συμβάλλουμε στην οικονομική μεγέθυνση. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που προωθούμε είναι απλούστευση των προγραμμάτων δαπανών. Συνεχώς μας λένε ότι είναι περίπλοκοι οι κανόνες και λειτουργούν ως αντικίνητρο για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες. Ανταποκρινόμενη λοιπόν σε αυτό η Κομισιόν προτείνει ριζική απλούστευση στο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, ε, ζητάει και από τα άλλα όργανα και τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειές της. Ας είμαστε ειλικρινείς. Θεωρητικά όλοι είναι υπέρ της απλούστευσης. Κανένας δεν έχει προτείνει ε, περαιτέρω περιπλοκή, αν θέλετε. Αλλά όταν μπούμε στις λεπτομέρειες, πολύ συχνά ο καθένας θέλει να προσθέσει το δικό του κανόνα, δική του αρχή και αυτό είναι πολύ κακό, πολύ αρνητικό όχι μόνο για τον προϋπολογισμό αλλά και για την εικόνα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τον προϋπολογισμό μας. Και ε, ε, όλα αυτά καθιστούν ε, τα μέσα αυτά δυσνόητα. 120 απλουστεύσει προτείνουμε συνολικά στους κανόνες ε, που διέπουν τις μικρομεσαίες, τις πόλεις και τις περιφέρειες, τους φοιτητέ, τους ε, ερευνητέ, αλλά και ε, το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. Ζητάμε μείωση των προγραμμάτων, μεγαλύτερη συνάφεια και σαφήνεια των κανόνων, καλύτερου στόχου και δείκτες, ε, πιο απλουστευμένες ε, μορφές επιχορηγήσεων και ε, αποφασιστική και πιο ταχεία καταβολή των πληρωμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ετούντες και βοηθάνε ε, βεβαίω ε, και την προώθηση τη ευρωπαϊκή οικονομία και των θέσεων απασχόληση. Είναι θέμα αξιοπιστία. Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε ε, από κοντά και θα γίνεται ένα απολογισμό τακτικά μέσω του scoreboard μα. Τώρα, η ε, αξιοπιστία είναι κάτι πολύ σημαντικό και η διαφάνεια. Προτείνουμε ένα σύστημα ίδιων πόρων σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό μας. Έτσι ώστε να έχουμε ένα ε, γενικό, ε, διαφανές και βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης. Η πρότασή μας για τους ίδιους πόρους βασίζεται σε έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ένα εξυγχρονισμένο πόρο ΦΠΑ με πιο ε, δίκαιη κατανομή του αντικτύπου μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτό από κοινωνικής απόψεως είναι πιο σωστό και ε, μετακυλείται, αν θέλετε, το φορολογικό, η φορολογική επιβάρυνση από την απασχόληση προς άλλες μορφές δραστηριότητας που επιβαρύνουν λιγότερο την ανάπτυξη. Από κάποιους υπολογισμούς που κάναμε, είδαμε ότι θα μειωθεί η εθνική συνεισφορά με αυτόν τον τρόπο κατά το ίμιση, κατά 50% μάλιστα υπολογίσαμε ε, θα μειωθεί τώρα με αυτά τα νέα μέτρα η εθνική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό ε, Προϋπολογισμό. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί έχουμε εδώ και τον Επίτροπο τον κύριο Λεβαντόφσκι που ε, θα σας εξηγήσει ακριβώς τη λογική αυτών των προτάσεων. Οι η πόροι, όπω είπε και ο πρόεδρο Σούλς, δεν είναι μια νέα ιδέα. Η συνθήκη είναι σαφέστατη σε αυτό το σημείο. Η Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτείται από του ίδιου πόρου τη. Θα πρέπει τώρα να έχουμε το θάρρο να μεταρρυθμίσουμε αυτό το σύστημα που είναι επεπαλαιωμένο και ιδιαίτερα περίπλοκο. Το ομολογώ. Ε, συμμετείχα από διάφορε ε, θέσεις ε, και εκπροσωπώντας την κυβέρνησή μου αλλά και ως επίτροπος ε, σε διαπραγματεύσεις για δημοσιονομικά πλαίσια. Σε δύο συμμετείχα τουλάχιστον. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει τώρα όλη αυτή η λογική της νόμιμης αν θέλετε επιστροφής, αποζημίωσης. Ναι, εντάξει, τη στιγμή που σπανίζουν οι πόροι και που μετράει και κάθε ευρώ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν σπαταλούνται οι πόροι. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θεσμικά όργανα και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν, που υλοποιούν τον ε, προϋπολογισμό. Και όπου είναι αδύναμη η φορείς θα πρέπει να ε, παρέχουμε εμείς κάποια ηχέγγυα και να αναλαμβάνουμε δράση. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό και το θέμα των υπερβολικών ελλημάτων. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος είναι μια διαδικασία που είχε συμφωνηθεί από όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνεπή τρόπο, ε, με ίστατο ε, σκοπό αν θέλετε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία αλλά και να ε, δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και οικονομική μεγέθυνση. Βλέποντας τώρα τα επόμενα βήματα, βλέπω ότι πολύ καλό προπαρασκευαστικό έργο γίνεται επί προεδρία Προεδρία σε τομεακό επίπεδο. Η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με την Προεδρία για την προετοιμασία των ε, ε, θεμάτων διαπραγμάτευσης και ευχαριστώ την Πρωθυπουργό, την Θόρνινγκ Σμιτ, για την προσωπική της δέσμευση στην όλη διαδικασία. Και καλωσορίζω τις παρατηρήσεις ε, που έκανε μόλις τώρα για αυτή την δέσμευση που εκφράζει για να συνεργαστεί μαζί μας αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι είναι μεγάλη η αφοσίωσή της, ε, γι' αυτό πιστεύω ότι ε, ναι, τα όργανα θα πρέπει να είναι αποφασιστικά βέβαια, αλλά και ευγενικά μεταξύ τους. Ε, προσβλέπουμε λοιπόν στην αγαστή συνεργασία και με το Συμβούλιο ε, και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον ε, κύριο Βαν Ρομπέι, εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και η δέσμευση των κρατών μελών μας ενδιαφέρει, αλλά και η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να προωθήσουμε τις συζητήσει μας έχοντας ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας όταν διαπραγματευόμαστε και εγκρίνουμε αυτή την δέσμη. Είναι γνωστή και η προσωπική και αφοσίωση του Προέδρου του κ. Σούλτ και τον ευχαριστώ για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην ενημερώνεται μόνο εκ των υστέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται εξ άντε, εκ των προτέρων η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχουμε μια πραγματική, σοβαρή, επικοδομητική διαπραγμάτευση. Χαίρομαι που έγινε ευρέω αποδεκτή η πρόταση τη Κομισιόν ω μια στέρεα βάση για τι διαπραγματεύσει ακόμη και από εκείνου που δεν έδειξαν και μεγάλο ενθουσιασμό για την πρότασή μα, θεωρούν παρόλα αυτά ότι είναι μια αξιόπιστη, στέρεα βάση για τι διαπραγματεύσει. Μέσα στου επόμενου μήνε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό ο προπολογισμό θα είναι ένα εργαλείο για να επενδύσουμε σε μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Ότι θα είναι ένα προπολογισμό που θα ε, είναι για όλου, για κάθε έναν από του Ευρωπαίου πολίτε μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Μπαρόζο, κυρία Πρωθυπουργέ. Μετά τις τρεις ομιλίες που ακούσατε τώρα, δεν ξέρω, ενδεχομένως να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα ή... Ευχαριστώ πάντως για την προσοχή σας. Έχει ανοίξει επίσημα η συνδιάσκεψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τόνα Σμιτ, τον κύριο Βαρόζο και καλή επιτυχία στις συζητήσεις σας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να καθίσετε να αρχίσουμε με το πρώτο πάνελ. Κύριε Μαυρογιάννη, κύριε Άνσεν, αν θέλετε να έρθετε στο Προεδρείο. Please take your seats. Σας παρακαλώ καθίστε. Θα αρχίσουμε. Αν θέλετε να καθίσετε και με την άδειά σας να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε με ε, το πρώτο τμήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε ε, τρεις ε, ε βασικές ομιλίες από τους τρεις ε, Είχαμε μάλλον τις τρεις, ε, τις ομιλίε ομιλίες από του τρει προέδρους και τώρα περνάμε στο πρώτο τμήμα. Είναι η δεύτερη συνδιάσκεψη για, τα, για το πολιετέ ε, πλαίσιο και για του ίδιου πόρους. Ξέρετε ότι ήδη υπήρξε μια πρώτη συνδιάσκεψη η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους με τους ε, ίδιους πρωταγωνιστές σε γενικές γραμμές. Πρόκειται σε μια, για μια συνδιάσκεψη που διεξάγεται στα ίδια πλαίσια και την ίδια χρονική στιγμή που ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα όργανα. Μια συνδιάσκεψη λοιπόν η οποία πιστεύουμε ότι θα χρησιμεύσει ιδιαίτερα για τις διαπραγματεύσεις αυτές για να ακουστούν τα επιχειρήματα των ΜΕ και των ΔΕ αλλά και για ε, να καταλάβουν οι πολίτες ε, που εκπροσωπείτε ποιες είναι οι απόψεις σας. Έχουμε 42 ε, μέλη εθνικών κοινοβουλίων που εκπροσωπούν 21 κράτη-μέλη. Έχουμε πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί μας και εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των άλλων θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία ε, θα λάβει χώρα ε, σε δύο τμήματα. Πρώτα απ' όλα θα ασχοληθούμε για τα έσοδα και για τους ίδιους πόρους και στη συνέχεια το απόγευμα θα ασχοληθούμε τις δαπάνες. Ακολουθούμε λοιπόν τους κανόνες της λογικής. Πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για τα έσοδα για να μιλήσουμε αργότερα και για τα έξοδα. Η συζήτηση αυτή ε, σίγουρα ε, θα ε, διεξαχθεί γύρω από τους κανόνες, ε, τους αριθμούς αλλά και τις πολιτικές και τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσεχή έτη. Μέσα σε ένα χρόνο περίπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάσει τον πρώτο προπολογισμό ε, του ε, πολιτικού πλαισίου 2014-2020. Ε, αυτές λοιπόν είναι κάποιες τεχνικής φύσει πληροφορίες και έχετε μπροστά σας αυτό το έγγραφο, αυτό το βελτίο. Είναι ένα βελτίο το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί να το συμπληρώσετε λοιπόν αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Να αναφέρετε το όνομά σας και το όργανο που εκπροσωπείτε. Τη χώρα σας, αλλά να μας πείτε εάν θέλετε να πάρετε το λόγο σήμερα το πρωί για τη συζήτηση επί των εσόδων ή το απόγευμα για τη συζήτηση επί των εξόδων. Μπορείτε βεβαίω να, να, μιλήσετε και το πρωί, να, να συμπληρώσετε και τα, τις δύο, και τα δύο τετραγωνίδια και, το πρωί και, για το πρωί και για το απόγευμα. Θα δούμε όμω, ε, γιατί πρέπει να κρατήσουμε και μια πειθαρχία όσον αφορά το χρόνο. Και θα δώσουμε βέβαια στο απόγευμα προτεραιότητα ε, στους, στα μέλη της διάσκεψης που δεν, θα έχουν που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν το πρωί. Ε, οι κλητήρε ε, ε, θα περάσουν κάποια στιγμή, όσο θα μιλούν τα μέλη του πάνελ, θα περάσουν να πάρουν τα βελτία αυτά τα οποία θα έχετε συμπληρώσει. Όπως πάντα, ως ήθιστε, στι συνεδριάσει που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να ακολουθήσουμε μια αυστηρή πειθαρχία όσον αφορά το χρόνο ομιλία. Μου ζητήθηκε να είμαι φιλικό αλλά και αυστηρό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι και τα δύο ταυτόχρονα. Μερικέ φορέ είναι κάπω δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω. Όσον αφορά ε, τι ομιλίε των μελών τη συνδιάσκεψη, ο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σα είναι δύο λεπτά. Σα παρακαλώ λοιπόν να ε, σεβαστείτε το χρόνο αυτό. Και τέλο, θα ήθελα να σα πω ότι οι εργασίες της συνδιάσκεψης στο σύνολό τους ε, μεταδίδονται διαμέσου του διαδικτύου. Οι πολίτες λοιπόν διαμέσου ε, ε, του δικτυακού τόπου του Κοινοβουλίου μπορούν να ακούν τις εργασίες μας και μέσω του Europe by Satellite να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά τις εργασίες. Ο καφές σερβίρεται έξω από την αίθουσα. Σας παρακαλώ για λόγους ευγένεια, αν θέλετε, να πάρετε τον καφέ σας έξω από την αίθουσα και να μην τον φέρνετε μέσα στην αίθουσα. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ, με την συμμετοχή του κυρίου Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι αναπληρωματής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από την Κύπρο εκφράζει ε, ε, τις τρεις προεδρίες του Συμβουλίου. Έχουμε την κυρία Εύα Κίαρ Χάνσεν, πρόεδρο της ε, ε Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ε, Κοινοβουλίου της Δανίας, εκπροσωπεί τα Εθνικά Κοινοβούλια, τον κύριο Ρεβαντόφσκι, επίτροπο, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Αν Τζένσεν, συν για τους ίδιους πόρους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία ε, εκπροσωπεί και τον κύριο Jean-Luc Dehaene, ο οποίος είναι ο δεύτερος συνεισηγητής του Κοινοβουλίου. Θα έρθει ε, σε λίγο η συγκήτρια του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Λεβαντόφσκι να μιλήσει εξ ονόμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στα εκλεγμένα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων 21 ε, χωρών. Πιστεύω ότι παρευρίσκεται ε, και την προσωπία της Κροατίας. Να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε με τα έσοδα. Εδώ και 20 χρόνια δεν συζητούσαμε ε, ή συζητούσαμε πολύ επιφανειακά το ζήτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή τώρα θέλουμε να προτείνουμε επαναστατικές θα έλεγα αλλαγές ε, όσον αφορά τα έσοδα. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση PowerPoint. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε μερικές φορές τη συνθήκη και να μην την ξεχνάμε. Ε, ήδη το έπραξε ο πρόεδρος Σούλτς. Μιλώ για το περίφημο άρθρο 311 της συνθήκης που αναφέρει αυτά τα οποία μπορείτε να διαβάσετε ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται πλήρως από τους ιδίους πόρους. Αυτό δεν είναι μόνο το πνεύμα, αλλά και το γράμμα της συνθήκης. Και ακριβώς γι' αυτό είπα ότι αξίζει το κόπο μερικές φορές να θυμόμαστε και τη συνθήκη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Και ε, μέχρι το 2011 η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική από το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης. Βλέπετε την... Βλέπετε την εξέλιξη ε, της συνιστώσας των εσόδων από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ε, στη δεκαετία του 70 έχουμε το πράσινο χρώμα, έχουμε ε, τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους, ε, τελωνία κυρίως, αλλά ήταν τότε μικρή κοινότητα και μικρό ο προπολογισμό. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 80, βλέπετε την μπλε ε, ζώνη ε, με το ΦΠΑ, αλλά τεχνητός υπολογισμός του ΦΠΑ. που αντικατέστησε πλήρως γύρω αντικαταστάθηκε πλήρως ε, στη δεκαετία του 90 από ε, τη βάση ε, του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Από την εποχή Σόιμπλε και Ροστόφκι και την εποχή τη δική μου βεβαίως, πιο μετριοπαθή στη συμβολή μου. Αυτή είναι η ιστορία της δεκαετίας του 90 όπου κυριαρχεί η βάση εθνικού ακαθάριστου εισοδήματος. Βλέπετε ότι εδώ μιλάμε για πραγματικούς προπολογισμού, για προπολογισμού που ψηφίζονται ε, και μάλιστα ε, για ε, προπολογισμού που έχουν εκτελεστεί. Βλέπουμε τη γενεοδορία με πάνω από το 1% του πραγματικού προπολογισμού, ενώ τώρα μιλάμε για πραγματικές δαπάνες μέχρι το 2011 στην Ευρώπη και για το γεγονό ότι είμαστε κάτω από το 1%. Και εδώ φτάνουμε σε αυτό το οποίο προτάθηκε τον Ιούνιο του 2011, αυτή τη σοβαρή αλλαγή που προτάθηκε στο σύστημα αυτό. Να σταματήσουμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε το στατιστικό ΦΠΑ από το 2014 και να έχουμε δύο νέους ίδιους πόρους. Ο ένας που να στηρίζεται στο ΦΠΑ και το άλλο ο φόρος επί των χρηματιστοτικών συναλλαγών. Και οι δύο επιλέγησαν από ένα μακροχελή κατάλογο υποψηφιωτήτων, αλλά μετά από μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγηση αντικτύπου, ε, υπήρξε αυτή η πρόταση για τους δύο αυτούς ίδιους πόρους. Και αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με ριζική τροποποίηση των λεγόμενων διορθώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο διαφανές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ΦΠΑ, που είναι ο ήρωα τη σημερινή μα. Ε, ε, και θα πάμε στον πραγματικό ήρωα τη σημερινή μα παρουσίαση, που είναι ο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εδώ μιλάμε για, ένα, ε, για το ΦΠΑ που είναι περισσότερο εναρμονισμένο, γι' αυτό και επελέγει, ω μέρο τη προσπάθεια να είναι πιο αποτελεσματικό στα πλαίσια τη ενιαία αγορά το σύστημα ΦΠΑ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. σω λοιπόν είναι ένα από του φόρου που πραγματικά προσφέρει Η μεταχείριση στα κράτη-μέλη. Η πρόταση λοιπόν στην ουσία τη, και πάμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι να ξεκινήσουμε αμέσως. Εδώ δεν υπάρχουν δυσκολίες στην συγκέντρωση και στον ε, υπολογισμό. Η πρότασή μας ήταν μέγιστο ποσοστό 2%, αλλά όσον αφορά την ε, εφαρμογή, ε, λειτουργικό ποσοστό, μιλάμε για 1% ε, της συγκέντρωσης των εσόδων με ε, ε, ε την ε, στάνταρ βάση. Τώρα έχουμε, αυτά όσον αφορά το ΦΠΑ, τώρα έχουμε δεύτερο υποψήφιο τον φόρο αυτό επί των συναλλαγών. Υπάρχει ήδη σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετική μορφή. Θέλαμε λοιπόν να διευρύνουμε την εφαρμογή αυτή. Κοιτάξτε, ε, να σας πω ότι ε, αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά παρουσιάζουμε ε, το κείμενο αυτό. Μιλάμε για ευρεία βάση, όχι μόνο για τις μετοχές, αλλά και για τα παράγωγα. 0,01 ε, για τα ε, παράγωγα και 0,1% ε, του, του συνολικού όγκου των τίτλων. Και ξεκινάμε ω εξή για τον υπολογισμό. Τα 2 τρίτα θα πάνε στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το 1 τρίτο το κρατούν τα κράτη-μέλη ω νέο πόρο των εθνικών προπολογισμών. Δεν θα επισέλθω τώρα στις λεπτομέρειες ε, όσον αφορά το σκεπτικό και την επιχειρηματολογία, αλλά πραγματικά ξέρουμε το πόσο οι φορολογούμενοι της Ευρώπης συμβάλλουν ε, στα διάφορα πακέτα διάσωσης ε, και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο δημοσιονομικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι εμείς Πιστεύουμε ότι καλύτερο να έχουμε έναν εναρμονισμένο ε, τέτοιο φόρο και σα είπα ότι υπάρχουν ήδη 10 κρατημέλη που εφαρμόζουν διαφοροποιημένο τέτοιο φόρο. Καλύτερα όμω ε, να ε, Καλύτερα να τον είχαμε σε παγκόσμια βάση αυτό τον εναρμονισμένο φόρο. Ξεκινάμε του 27. Πάντω ε, εδώ δεν θα αυξηθούν οι δαπάνες, αλλά εν μέρη θα υποκαταστήσουν ε, τις εθνικές δαπάνες και τις εθνικές συνεισφορές. Και ο πρόεδρος Μπαρόζο το είπε. Ε, η φορολόγηση από την εργασία θα μεταφερθεί στο κεφάλαιο και θα ανταμείβονται οι μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και επενδύσεις. Γιατί εδώ μιλάμε για τη φορολόγηση των συναλλαγών. Και κυρίως των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών η αρχική βάση για τους υπολογισμούς ε, ε, ε, έχει ως εξής. Υπολογίζουμε 57 περίπου δις, άντληση 57 δις κατά προσέγγιση, με την προϋπόθεση ότι φορολογούνται και τα δύο μέρη της συναλλαγής. Όταν, μια, όταν ένας γαλλικός θεσμός, και μιλούμε για θεσμούς, έτσι, το 85% ε, ε, ε, των συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αλλαγές αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, όλους, όλα τα ταμεία ε, συλλογικής αποταμίευσης, ε, συνταξιωτικά ταμεία κτλ. Δεν μιλάμε για νοικοκυριά ή για δάνεια, μιλάμε για θεσμούς. Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα ενός γαλλικού θεσμού που διαμέσου της Φραγκφούρτης διαπραγματεύεται με ένα σουηδικό θεσμό Ε, ε, κοιτάξτε, η εισπράξη θα γίνει και στη Γαλλία και στη Σουηδία. Εμείς υπολογίζουμε για το 2010 τις εκτιμήσεις μας με βάση ε, τα τα ευρω... τη συνομοσπονδία των ε, Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Τίτλων και από την, ε, τα κεντρικά γραφεία συμψηφισμού. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με, την με το παράδειγμά μας αυτό, με αυτή την προϋπόθεση και, έχουμε κάνει μια πρόβλεψη των εξελίξεων. Μην ξεχνάμε ότι το 2010 στηρίζεται σε πραγματικά στατιστικά στοιχεία. Με την προπόθεση όμω ότι ε, αυτό ο φόρο θα μπορούσε να έχει επιπτώσει στου όγκου, ήδη έχουμε μειώσει τη βάση για το 2010 για τα εισοδήματα κατά 70% για τα παράγωγα. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει επίπτωση στο εμπόριο στι συναλλαγέ, κυρίω όσον αφορά τα πιο εξελιγμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα παράγωγα, ενώ πολύ μικρότερο πολύ μικρότερος είναι ο αντίκτυπο στι μετοχέ και στα ομόλογα. Αυτή είναι η βάση υπολογισμού. 38 που θα συγκεντρωθούν το 2010. για τον ευρωπαϊκό, ε, υπολογισμό, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. και 54 για το, για το επόμενο έτος. Γιατί είπαμε ότι το 1 τρίτο πάει στου εθνικού προπολογισμού. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι φορολογούνται και οι δύο πλευρές της συναλλαγής. για όλα τα ιδρύματα τα οποία είναι καταχωρημένα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε τις, ε, τις προβλέψεις μας ήταν πιο αισιόδοξε έναντι του Ιουνίου σε σχέση με τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε ως μείωση της συνεισφοράς ε, στον προπολογισμό των κρατών μελών. Βλέπετε εδώ. Η πρώτη στήλη είναι η συμβολή εθνικού ακαθάριστου ε, Γερμανίας, Γαλλίας και των άλλων πρωτευουσών και το, πώς να το πω, το γαλάζιο, το τυρκουάζ, η επόμενη στήλη. Αφορά τη συνεισφορά των κρατών μελών, λαμβάνοντα υπόψη τον φόρο. Για παράδειγμα, για την Ολλανδία, 2,6 δις ευρώ μείωση τη εθνική συνεισφορά θα μπορούσαμε να έχουμε. 1,8 για την Πολωνία, 1,8 δις. Και το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε και για τι μικρότερε χώρε ή του καθαρού ε, ε, δικαιούχου και τελικό ε, γράφημα είναι ε, προβλέψη μέχρι το 2020. Ε, ο φόρος αυτός θα υποκαταστήσει λοιπόν τη βάση του ΑΕΠ. Και έχουμε και, το, και την κατάσταση του παλιού περίπλοκου συστήματος ΦΠΑ με το καινούριο. Δεν έχω τον καιρό να σας αναφέρω την πρότασή μας για τους μηχανισμούς διόρθωσης. Έχουμε νέε διορθώσει ε, και εδώ είμαι έτοιμο ε, ε, να σα αναφέρω την πρότασή μα όταν θα γίνει συζήτηση και οι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Commissioner, Lewandowski. Mr. Andreas... Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι. Ο κύριο Αντρέα Μαυρογιάννη, αναπληρωτή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τη Κύπρου, της Κύπρου εκπρόσωπος της Τριάδας των Προεδριών του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι ομιλητές, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, ε, θα ήθελα να εκφράσω εδώ την εκτίμησή μου ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Δανική ε, Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διοργανώνει αυτή τη δεύτερη διάσκεψη για το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης με έκδηλα αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία μας. Το επόμενο πολιετές πλαίσιο θα είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το μέλλον μας και η συζήτηση θα πρέπει να εστιαστεί γύρω από τις βασικές αρχές που στηρίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα και η διαφάνεια και γύρω από τους κοινούς μας στόχους και η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι απλώς παράθεση θέσεων. Θα πρέπει να πάμε πιο μακριά. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει σαν στόχο την οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτησή μας θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στις ανάγκες και στις φιλοδοξίες. Δεν θα πρέπει να είναι απλώς ε, μία συζήτηση για στοιχεία και ποσοστά. Οι αποφάσει για τους πόρους και τους μηχανισμούς ε, της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού ε, προπολογισμού είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορα οικονομικά κριτήρια όπως είναι η οικονομική αποδοτικότητα, η σταθερότητα και η επάρκεια. Διοικητικά επίση κριτήρια όπω είναι ε, η ή, πολιτικά ε, κριτήρια όπως είναι η σχέση με τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς. Η ε, χρηματοοικονομική αυτάρκεια, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, τώρα ουσιαστικά σχετίζεται με τη γενικότερη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ε, όπως μόλις τώρα υπενθύμησε η Πρωθυπουργό της Δανίας. Μία επίκριση αυτή τη στιγμή είναι ότι το νυν σύστημα δεν είναι διαφανές, δεν είναι σαφές. Πολλά έχουν ακουστεί και ο πρόεδρος Σούλτ μόλις μας υπενθύμησε και το άρθρο 311. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν ξέρουμε ουσιαστικά εάν μπορούμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι είναι ε, πραγματικά ίδιο σπόρος η εθνική συνεισφορά. Το ίδιο ισχύει και για το στατιστικό ΦΠΑ, που βασίζεται ουσιαστικά σε, μια εθνική συνεισφορά. Ως τέτοιο θεωρείται πολύ συχνά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι σε τελική ανάλυση το πραγματικό ερώτημα σήμερα δεν είναι αν χρειαζόμαστε ίδιους πόρους, αλλά ποιοι είναι οι καλύτεροι ίδιοι πόροι που μπορεί να έχουμε, σε ποια επίπεδα, με ποιες εφαρμοστικές λεπτομέρειες κτλ. Εξάλλου, στην καρδιά του θέματος βρίσκεται το ζήτημα μιας πολύ συγκεκριμένης δέσμευσης ώστε να παρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κατάλληλα οικονομικά μέσα που θα αντιστοιχούν στο επίπεδο των φιλοδοξιών μα. Και αυτού, του χαλεπού καιρού, ίσω περισσότερο παρά ποτέ, θα πρέπει να έχουμε υψηλέ προσδοκίε και φιλοδοξίε, και ε, ε, να βοηθήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να καλύψει τι ανεπάρκειες των εθνικών προπολογισμών. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και σε οικονομικού όρου είναι πολύ καλύτερο τα πράγματα να γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολλέ φορέ από ότι σε εθνικό υπογράμμισε και ο πρόεδρος Μπαρόσο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις της Κομισιόν, ένα ίδιο πόρο ΦΠΑ θα βασιστεί στην ίνη υποδομή ίσπραξη ε, του φόρου. Η εφαρμογή θα είναι πιο εύκολη από ό,τι άλλε επιλογέ. Θα παράσχει ε, σταθερή ε, και σταθερά έσοδα με το ελάχιστο διοικητικό κόστο. Ενώ έτσι οι πολίτε μα θα ξέρουν καλύτερα πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Από την άλλη πλευρά όμω αναγνωρίζεται ότι ένα ίδιο πόρο ΦΠΑ θα παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα προβλήματα ανισότητας που υπάρχουν τώρα στα εθνικά συστήματα και ε, επιβάλλει περισσότερες επιβαρύνσεις στα κράτη-μέλη ε, που έχουν ε, το υψηλότερο μερίδιο, αν θέλετε, στην οικονομική δραστηριότητα. Έτσι θα αυξηθεί η συνεισφορά κατά πολύ για ορισμένα κράτη-μέλη και όχι για τόσο, τόσο, κατά τόσο πολύ για άλλα κράτη-μέλη. Λαμβάνοντας τις νυν κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, θα μπορούσε η επιβολή ενό τέτοιου φόρου να αποξενώσει τους πολίτες. Η άλλη πρόταση αφορά ε, έναν φόρο για τι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Θα μπορούσε να παρέχει σημαντικά έσοδα χωρίς ε, ιδιαίτερη δυσκολία στην ίσπραξή του. Αυτός ο φόρος νομίζω ότι θα εκτιμηθεί από την πλειονότητα των, ε, πολιτών μας ε, δεδομένων των ε, νυν συνθήκων. Πολλοί βέβαια επιχειρηματούν και λένε ότι θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου που δεν έχουν επιβάλει αυτό το φόρο. Είναι ιδιαίτερα επίμαχο αυτό το θέμα, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν πολύ ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό τομέα και ε, χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα για να ορίσουν την φορολογική βάση. Η σταθερότητα εξάλλου του προπολογισμού ε, θα μπορούσε να επηρεαστεί από του οικονομικού κύκλου και θα είναι αβέβαιο αυτό το έσοδο και θα μπορούσε να οδηγήσει μάλιστα και σε μεγάλη μείωση των συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήγοντα την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού μα τομέα και ε, τη οικονομική μα δραστηριότητα. Εν, καιρό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει όμως για να αποφασίσουμε να εξετάσουμε και όλες τις άλλες εφαρμοστικές λεπτομέρειες, κυρίως το στοιχείο για την κατοικία, residence, που είναι τμήμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι ο πραγματικός οικονομικός και χρηματοπιστωτικός αντίκτυπος και όλες οι άλλες συνέπειες ε, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Ούτως ή άλλως εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότερες εξηγήσει και αποσαφηνήσεις σε αυτό το τομέα και πιο συγκεκριμένα. Αυτό που μόλις τώρα είπε ο Επίτροπος Λεβαντόμφσκι θα πρέπει να μας δώσουν τροφή για προβληματισμό. Μετά η Κομισιόν προτείνει επίσης ε, και ε, κάτι για του μηχανισμούς διορθωση. νέους μηχανισμούς διορθωση Είναι πολύ επίμαχο το θέμα των ε, διορθώσεων. Η εισαγωγή των καταποκοπήν ποσών θα αυξήσει την διαφάνεια και την ε, δικαιοσύνη. Σίγουρα εδώ θα πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές Φοντανεμπλό. Μπορεί κανεί να πει ότι ε, δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέλειο ίδιο πόρο. Η κάθε επιλογή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τη και θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά υπόψη την οικονομική και την πολιτική πραγματικότητα. Τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να έχουν διαφορετικές απόψεις ε, για τις διάφορες επιλογές. Η επάρκεια και η ε, δικαιοσύνη όμως είναι δύο αρχές που μας καθοδηγούν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επαρκείς φόρους. Ε, εσόδων και για την Κομισιόν και για το Κοινοβούλιο. Οι μεταρρυθμίσει είναι αλήθεια ότι κάνουν ε, πιο απλό το σύστημα των ίδιων πόρων. Δεν είναι όμως αυτό σίγουρο ότι θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε ε, προβλήματα όπως οι διορθώσεις που, ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το σκέλος δαπάνες του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε σε 20 δευτερόλεπτα, ε, παρόλο που καθυστέρησα, θα ήθελα να κλείσω με ένα θετικό τόνο. Είμαι πεπισμένος ότι η συζήτηση μεταξύ ημών εδώ σήμερα θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τα τέλη του έτους. Ξέρω ότι γι' αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και στο θέμα των ίδιων πόρων. Είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι απόψεις όλων των θεσμικών οργάνων. Αλλά θα πρέπει να βρούμε μια λύση λαμβάνοντας υπόψη τους ε, ε, χαλεπούς ε, καιρούς ε, μεν που θα μας βοηθήσει ε, δε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους Ευρώπης 2020. Υπό αυτή την έννοια η σημερινή διάσκεψη μας δίνει μια θαυμάσια ευκαιρία για μια ε, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κοντά ήσασταν πάνω στο χρονικό όριο. Η κυρία Εύα Κερ Χάντσερ, πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δανίας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Είναι αρκετά σπάνιο να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θεμελιώδη ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζω αυτή τη συζήτηση αν και δεν είναι το πιο εύκολο θέμα να αντιμετωπίσουμε, ιδίως, και ιδίως δεν είναι το πιο εύκολο ζήτημα σε έναν καιρό, σε μια εποχή που τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ε, σκληρούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό. Είχαμε μια συζήτηση τη Δευτέρα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο σε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση στην, ε, στην Κοπενχάγη. Και ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξαν πολλέ διαφορετικέ απόψει για το πώ να δαπανηθούν χρήματα, ιδιαίτερα εν καιρό κρίση. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι ζωτική σημασία η Ένωση να βασίζεται στι αρχέ τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Αν θέλει να, τη, να την χάνει τη υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτέ οι αρχέ πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσει η Ένωση, αλλά και στι συγκεκριμένε πολιτικέ. Και γι' αυτό και στην πλευρά των εσόδων της, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Τώρα θα ήθελα προσπαθήσω να εκτιμήσω, την, ε, να αξιολογήσω την πρώτη επιτροπή για τα έσοδα για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με βάση αυτές τις αρχές. Όπως μόλις ακούσαμε υπάρχουν δύο νέοι ήδη υπόλοιποι που προτείνω την Επιτροπή. Αλλά προτού σχολιάσω αυτές τις δύο προτάσεις θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Νέοι ήδη υπόροι. Εκτός του ότι πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς, πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια. Πρώτα απ' όλα η πλειονότητα στο Συμβούλιο πιστεύει ότι η ίσπραξη των φόρων πρέπει να παραμείνει μια εθνική αρμοδιότητα. Πρέπει να είναι θέμα των εθνικών κοινοβουλίων να αποφασίσουν ποιοι, φόροι εισπράττονται. Δεύτερον, τα έσοδα και τα επιτόκια από, από του ίδιου πόρου θα πρέπει να αποφασίζονται είτε από το να αποφασίζονται μόνο από το Συμβούλιο που αντιπροσωπεύει τις θέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είναι ρεαλιστικό να, να οραματιστούμε εδώ μια διαφορετική προσέγγιση. Και τρίτον, τα έσοδα από τους νέους ίδιους σπόρους πρέπει να οδηγήσουν σε μια μείωση της συνεισφοράς ε, στο, του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών. Οι νέοι ίδιοι πόροι δεν πρέπει να είναι ένα τρόπο για να αυξηθεί το γενικότερο επίπεδο εξόδων στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τώρα να πω λίγα λόγια για το νέο ίδιο πόρο ΦΠΑ. Ο στόχο τη Επιτροπή είναι να απλοποιήσει το, τον, υπολο, τον υπολογισμό του ΦΠΑ και να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών. Αυτό ταιριάζει καλά με τα κριτήρια της δικαιοσύνης και διαφάνειας που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου. Αλλά η ανησυχία μου είναι αυτή τη στιγμή ότι οι επιπτώσεις για, τα, για τις συνεισφορές των διαφόρων κρατών μελών δεν είναι ξεκάθαρες. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι πιθανό να υπάρχει μια εκτίμηση του κατά πόσο ο, ο, ο ίδιος πόρος του ΦΠΑ οδηγεί σε ένα σε έναν ισότιμο καταμερισμό του βάρου μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό θα ήθελε η Επιτροπή να μα παρουσιάσει πληροφορίε σχετικέ με αυτό, όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Και τώρα λίγα λόγια για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η πρόταση για τον φόρο αυτό θέτει δύο ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει γενικά να υπάρχει ένα τέτοιο φόρο στην Ευρώπη. Και αυτή η ερώτηση από μόνη της είναι αντιφατική. Ε, και μετά, Ποιε είναι οι επιπτώσεις ενός τέτοιου φόρου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ανυπομονώ να μελετήσω σε λεπτομέρεια το, το νέο υπολογισμό που παρουσίασε η Επιτροπή για το πώς αυτό θα επηρεάσει τον ΑΕΠ της ε, Ένωσης και την ανεργία. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση. Και δεύτερον, αν υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη για ένα τέτοιο φόρο, τότε τα έσοδα θα βγουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή μόνο στου εθνικού προπολογισμού. Και εδώ χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε για τι επιπτώσει τη διανομή. Φαίνεται απίθανο η πρόταση της Επιτροπής να μπορέσει να, να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά για πολλές χώρες επίσης που είναι υπέρ του φόρου, Επιμένω αυτέ οι χώρε ότι τα έσοδα θα πρέπει να πάνε στα, στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς και όχι στον ενωσιακό. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στους μηχανισμούς διόρθωσης. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι γνωρίζετε από την εθνική πολιτική ότι αντιμετωπίζουμε παρόμοιες συζητήσεις όταν μιλάμε για μετάφορα πόρων μεταξύ περιοχών. Ποιος θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο, ποιος θα πρέπει να πληρώσει λιγότερο. Ο υπολογισμός πάντα γεννά συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Στην καλύτερη περίπτωση θα προτιμούσα να μην υπάρχουν διορθώσεις στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Αλλά τούτου λεχθέντος θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το ισχύον σύστημα διόρθωσης δεν είναι δίκαιο και δεν είναι μια βιώσιμη λύση τουλάχιστον κράτη-μέλη τα οποία είναι ισότιμα όσον αφορά το οικονομικό τους καθεστώς θα πρέπει να την χάνουν ισότιμης μεταχείρισης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε από τις χώρες που, που είναι τώρα δικαιούχοι του μηχανισμού διόρθωσης να μετακινηθούν στις, προ... στις θέσεις τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια καλύτερη λύση για τις διορθώσεις. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι κάθε φορά που έχουμε μια συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπάρχει μια υπάρχει αίτημα για περισσότερα χρήματα για νέου τομεί πολιτικής. Τι θα γίνει αν εμεί, αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίσουμε να μιλάμε για το πώς στην πράξη θα δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα. Ποια είναι, ποια είναι η επίπτωση των διαφόρων θέσεων στον προπολογισμό. Γνωρίζουμε πολλά για το τι αλλαγές θα επιφέρει στον τρόπο που δαπανούμε τα χρήματα σήμερα. Ενδεχομένω κάποια θα μπορούσαν να δαπανηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο και περισσότερα στα μελλοντικά κέρια ζητήματα για το πώς να έχουμε ενδεχομένω νέες επενδύσεις, μια πιο πράσινη Ευρώπη, περισσότερη ανάπτυξη κτλ. Ο Επίτροπος άρχισε λέγοντας ότι ο προπολογισμό θα χρηματοδοτηθεί και εμεί πρέπει να δούμε, να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επτά λεπτά. Ακριβώς. Και τώρα η κυρία Γένσεν, για τους ίδιους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και ευχαριστούμε που διοργανώσατε αυτή τη διάσκεψη που νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τα όσα είπε η κυρία Χένσεν. Πράγματι, οι νέοι ήδη πόροι θα πρέπει να σέβονται ε, την εθνική δημοσιονομική κυριαρχία. Και εμείς το πιστεύουμε. Τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά που θα πρέπει να αποφασίσουν τη φορολογία στην Ευρώπη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλουμε να το συζητήσουμε το ζήτημα μαζί σα. Δεύτερον, είπε ότι ε, τα έσοδα θα τα αποφασίσει το Συμβούλιο. Ναι, αλλά αφού ακούσει την άποψη του Κοινοβουλίου, θέλουμε να σα εμπνεύσουμε. Έχουμε λοιπόν ε, τη ε, διαδικασία αυτή τη ακρόαση. Και βεβαίω είναι αλήθεια ότι την απόφαση την παίρνει το Συμβούλιο. Τέλο, ακούσαμε ότι οι νέοι ήδη πόροι θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση τη εθνική συνεισφορά. Μα ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι και η δική μας άποψη. Αυτό ζητάμε. Μείωση των εθνικών συνεισφορών ε, με ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Γιατί θέλουμε αυτό το νέο σύστημα. Για να έχουμε ένα απλούστερο, διαφανέστερο και κατανοητό σύστημα ιδίων πόρων. Και εδώ λοιπόν συμφωνούμε με όλα αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία κερ Χάνσεν σε σχέση με το γεγονός ότι η λέξη κλειδιά είναι διαφάνεια και δικαιοσύνη. Ζητάμε λοιπόν οι νέοι ήδη πόροι ε, να αποτελέσουν προϋπόθεση για να συμφωνήσουμε και να υπερψηφίσουμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ έχουμε αρμοδιότητα. Πρέπει να συμφωνήσουμε, να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και είπαμε ότι αν δεν καταλήξετε σε ένα δικαιότερο, απλούστερο και πιο διαφανές σύστημα για τους ίδιους πόρους, μπορεί τελικά το Κοινοβούλιο να πει όχι στο ε, πλαίσιο. Και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η συνολική συζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και για τους ίδιους πόρους στην ουσία είναι πολύ δύσκολη. Ε, το ζήτημα είναι πολύ λεπτό και στο Συμβούλιο. Ε, εκεί πρέπει να πούμε ότι γίνεται ένα παζάρι ανάμεσα στου αρχηγού κρατών κυβερνήσεων. Και επιτρέψτε μου να σα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιε συζητήσει, ο επικεφαλή των συζητήσεων ε, εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τόνι Μπλερ, είπε την επόμενη φορά θα αλληλοσκοτωθούμε. Ε, δεν είναι και πολύ ωραία όλα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να μπορέσετε ε, ε, να δουλέψετε σε ένα καλύτερο κόσμο. Το κλίμα να είναι καλύτερο, οι συζητήσει να είναι καλύτερες, να εστιάσετε την προσοχή σας περισσότερο στις δαπάνες και λιγότερο στη δίκαιη επιστροφή να εστιάσετε την προσοχή σας στις ποιότητες. Γιατί και να μην κολλάτε στις δαπάνες όπου ο καθένας προσπαθεί να ε, αντλήσει περισσότερα ωφέλη και να είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση ένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ε, το, ε, τους δύο ε, νέου ίδιους πόρους, τον, το ΦΠΑ, τη βάση ΦΠΑ, τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αυτά συζητούνται και στα πλαίσια τη ιστορική αγορά, αλλά και στα πλαίσια των ιδίων πόρων. Πρέπει να σα πω ότι η σαφή, μου εντύπωση είναι ότι η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ε, συμφωνεί με αυτές τις υποδείξεις της Επιτροπής. Άρα, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ε, είναι, ε, συμφωνούν, συμβαδίζουν σε συγκεκριμένο σημείο. Εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Προπολογισμού συζητάμε αυτή τη στιγμή το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και σκεφτόμαστε το εξή. Εάν εσεί συμφωνήσετε σε αυτό το φόρο, τότε τουλάχιστον ένα τμήμα των εσόδων ε, θα προέρχεται από τους νέους ιδίους πόρους, άρα θα έχουμε μείωση της εθνικής συνεισφοράς. Και ε, πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένω, συνοψίζοντα, θέλω να είμαι πολύ σαφή σε αυτό το οποίο θέλουμε εμεί στο Κοινοβούλιο. Επιθυμούμε ένα πλούστερο σύστημα ιδίων πόρων, ένα σύστημα που να μην προβλέπονται εξαιρέσει και εκπτώσει. Όχι, δεν θέλουμε δηλαδή 42 εξαιρέσει που έχουμε στο παρόν σύστημα και από μεριά εσόδων και από μεριά δαπανών. Δεν θέλουμε υψηλότερους ε, ε, καθαρούς φόρους, υψηλότερους φόρους σε απόλυτες τιμές. Θέλουμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των ιδίων πόρων. Θέλουμε να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ποιότητα των δαπανών, ε, στο σκέλος δαπάνες. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε κατά την άποψή μας. Στον ευρωπαϊκό υπολογισμό δεν θέλουμε δαπάνες που να ωφελούν μόνο την καθαρή θέση ορισμένων χωρών οι δαπάνες υφίστανται διότι είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την εσωτερική αγορά, για την συνοχή ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε να μειωθούν οι εθνικές σας συνεισφορές. Μα αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν να το ακούσατε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τώρα με τις παρεμβάσεις ε, από την αίθουσα. Ε, ελπίζω να συμπληρώσετε όλοι το έντυπο. Διαφορετικά σηκώστε το χέρι σας και θα σας σημειώσουμε. Δίνουμε πρώτο λόγο στον κύριο Εδουάρδο Καμπρίτα, πρόεδρο ε, της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την πρωτοβουλία ε, που πήρατε να γίνει αυτή η συζήτηση, αυτή η ανοιχτή συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ε, θελήσατε να συμμετάσχουν και τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι ε, σήμερα ε, οι συνθήκες ε, που επικρατούν είναι πιο ευνοϊκές από το κλίμα το οποίο επικράτησε στην πρώτη συνδιάσκεψη το θέμα αυτό το φθινόπωρο. Σήμερα ε, τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά πλαίσια ε, είναι καλύτερα, είναι πιο σταθερά και ε, έχουμε προχωρήσει περισσότερο στην εργασία μας έτσι ώστε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να είναι ένας προϋπολογισμός που να προωθεί την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη που τη θέλουμε όλοι να είναι πιο ανταγωνιστική. Και γι' αυτό η συζήτηση για τους ίδιους πόρους θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής απάντησης, κοινή απάντησης, απέναντι σε μια κρίση η οποία ε, η κρίση δεν αφορά το α ή το β ε, κράτος μέλος συγκεκριμένα. Είναι μια ε, συνολική κρίση, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, αφορά ιδιαίτερα ε, την ε, ζώνη του ευρώ ε, και βεβαίως την κρίση αυτή τη ζει με διαφορετική ένταση κάθε χώρα. Σε αυτά τα πλαίσια, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να προωθεί την αλληλεγγύη, την ανταγωνιστικότητα και την ισορροπημένη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκά πλαίσια με βάση όλα αυτά, οι νέοι ήδη πόροι θα πρέπει να ενισχύσουν αυτή την ιδέα της δικαιοσύνης ως προς την ε, κατανομή της χρηματοδότησης ε, στα, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χρονικό διάστημα 2014-2020. Και όσον αφορά ε, το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, εδώ ε, θα πρέπει να πούμε ότι ο φόρος αυτός ανταποκρίνεται ε, στην απέτηση να υπάρξει μια συνένεση που να επιτρέπει από τη μια να εφαρμόζουμε τη συνθήκη, δηλαδή να χρηματοδοτούμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό κυρίως από τους ίδιους πόρους. Ταυτόχρονα όμως θα επιτρέψει να δοθεί μια απάντηση στους Ευρωπαίους πολίτες σε σχέση και να δοθεί η απάντηση έναντι των Ευρωπαϊκών πολιτών σε αυτή τη συνολική κρίση. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα να χαρακτηρίζεται από ισορροπία ε, και να χρηματοδοτεί τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και ε, με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και αυτή η μείωση των εθνικών συνεισφορών. Ε, σύμφωνα με το εθνικό ακαθάριστο εισόδημα κάθε κράτου μέλου. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μα προ την κατεύθυνση αυτή. Σε εμά, στη χώρα μα, υπάρχει σε ιστορικό επίπεδο ευρεία συνένεση. θα πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση βεβαίω, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί προτεραιότητα στι επενδύσει που θα προωθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Mr. Ludek Chair of the European Union Affairs Committee in the Senate of the Czech Republic, Ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, της ε, Τσεχίας ε, για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω ένα σχόλιο. Όταν προετοιμάζαμε την Προεδρία μας, το πρώτο εξάμεινο του 2009, είχαμε την εντύπωση ότι τότε θα γινόταν η ενδιάμεση ε, αξιολόγηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Και ε, πραγματικά εξεπλάγημεν όλοι όταν είδαμε ότι αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση έγινε δύο χρόνια μετά. Αυτό δεν ε, είναι μια επίκριση, απλώς μια προειδοποίηση. Διότι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ ε, αξίζει τον κόπο να γίνει και αξίζει τον κόπο να αντλήσουμε κάποια μαθήματα. Εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ξεκίνησαν εγκαίρως ε, τώρα τη συζήτηση και το θέμα συζητήθηκε και ε, στην ε, Τσεχία, στη Γερουσία. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ της πρότασης Ε, για απόσυρση όλων των μηχανισμών rebate. Είπατε ότι δεν θα στοιχήσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω προπολογισμό. Τέλειο αυτό σε αυτές τις συνθήκες κρίσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ε, κατάσταση ε, στην οποία ζουν οι συμπολίτες μας και δεν μπορούμε να τους υποσχόμαστε τίποτα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει μία προστιθέμενη αξία. Οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να συνδεθούν με αυτό, με το ότι θα επιφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία ε, οι πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να ωφελήσει τους πολίτες ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. χωρίς να απορροφήσει περισσότερα κονδύλια που χρειάζονται σε εθνικό επίπεδο για συντάξει και για οτιδήποτε άλλο. Εμείς ε, τώρα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε και να αξιολογήσουμε τις υπόλοιπες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Euh, Το λόγο έχει η κυρία Περβάν Μπέρες. Ευχαριστώ. Ε, euh, Θα ήθελα ε, και εγώ να ε, συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για του ίδιου πόρου. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή τη κρίση, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι τέτοια που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε την πηγή έμπνευση των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ακριβώς ε, ήδη από τότε είχε ξεκινήσει αυτή η ανάπτυξη των ιδίων πόρων και αυτό φάνηκε από το γράφημα που δείξατε στα πλαίσια αυτού του πνεύματος και λαμβάνοντας υπόψη ε, και, τη, και τη νέα διάσταση στις συνθήκες όσον αφορά τον ορισμό των ιδίων πόρων, νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ισορροπία. Γιατί το να ορίσουμε ε, ένα ίδιο πόρο ή ένα φόρο, σε κάθε οικονομία πρέπει να καλύπτονται οι εξή στόχοι. Πρώτα απ' όλα, να υπάρξουν οι πόροι έτσι ώστε η να υπάρχει χρηματοδότηση ε, από... Ε, σε δημόσιο επίπεδο. Δεύτερον, ε, δίκαιη κατανομή ανάμεσα στους πολίτες και στους φορολογούμενους, αλλά ταυτόχρονα να παροτρύνονται οι οικονομικοί πρωταγωνιστές προς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και βεβαίως πρέπει να τα πολιτεύσουμε όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι αυτά που προτείνεται ανταποκρίνονται απόλυτα σε αυτούς του τρεις στόχους. Πιστεύω ότι ε, εμείς πρέπει να σκεφτούμε αυτό τον ειδικό φόρο στα πλαίσια αυτής της ισορροπίας, όπου φαίνεται ότι όλοι έχουν συμφέρον. Δύο τρίτα Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα τρίτο τα κράτη-μέλη, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι ενισχυμένη συνεργασία ορισμένων κρατών μελών. Όχι, θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, διαφορετικά, ε, εάν στόχο είναι μόνο οι πόροι ε, για τα κράτη-μέλη, θα χάσουν το ενδιαφέρον τους οι υπόλοιποι. Γιατί εδώ μιλάμε κατά κάποιο τρόπο για το ΦΠΑ του 21ου αιώνα. Αυτόν ε, που στηρίζεται στην ανάπτυξη μια δραστηριότητα που μέχρι στιγμή διέφυγε από κάθε μορφή σε φορολογία. Και τέλο, Θέλω να επανέλθω σε αυτήν την ιδέα ότι διαμέσου τη φορολογία των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, με την ε, αντίστοιχη ισορροπία από τον, από τον πόρο ΦΠΑ θα έχουμε δικαιοσύνη έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Μα αυτό είναι απόλυτα σημαντικό κατά την άποψή μου. Κυρίω γιατί, ε, όπω είπαμε, ένα τρίτο θα ωφεληθούν τα κράτη-μέλη. πολύ σημαντικό. θα έχουν συμφέρον λοιπόν και τα κράτη-μέλη γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η εθνική συνεισφορά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριος Πιέρ ε, Μπερνάρ, μέλος της Γαλλικής Γερουσίας. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη θα συνεχίσει να δείχνει ασήμαντη στον κόσμο με έναν προϋπολογισμό που αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΚΠ. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι μόνο μία λέσχη λίγων που περνάει το χρόνο της μιλώντας για μείωση των συνεισφορών, προωθώντας αυτή την ε, οδηγή, τη θεωρία της δίκαιης επιστροφής ε, και συζητώντας για τα rebates, για τις εκτόσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει τις αυστηρές ε, πολιτικές. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να υποχωρήσει αλλά να προωθήσει ε, τα σχέδιά της για τις πολιτικές ανάκαμψης ε, και ανάπτυξης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα μας επιτρέψει να δούμε αν η Ευρώπη μπορεί να αναδυθεί από τις τάχτες της. Ε, είναι Πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα. Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού μέχρι το 2020 που θα αντιπροσωπεύει τότε το 2% ε, του ΑΕΚΠ. Ε, το να ελαφρύνουμε τις συνεισφορές ε, του κάθε κράτους. Πράγμα που θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό το περιθώριο αν θέλετε σε ό,τι αφορά τη μείωση του δημόσιου χρέους. Το να δώσουμε την ευκαιρία στην Ευρώπη να αποκτήσει ένα πιο συνεπή προϋπολογισμό. Αυτοί οι τρεις στόχοι δεν θα επιτευχθούν παρά μόνο εάν οι ίδιοι οι πόροι που αντιπροσωπεύουν τώρα το 14% του προϋπολογισμού φτάσουν στο 60% περίπου μέχρι το 2020. Αυτό προϋποθέτει ότι θα υιοθετηθούν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ίδιος πόρος για το ΦΠΑ και ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε που θα μπορούσε ακόμη να προσαρμοστεί περαιτέρω. Αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλους ίδιους πόρους που θα μπορούσαν να έρθουν να προσθεθούν στους δύο πρώτους ή να αντικαταστήσουν κάποιον από αυτούς εάν αποτύχουν. Ο φόρος επί του καπνού ε, και τα ινοπνευματόδη για παράδειγμα ή ε, ένα τμήμα, ε, μια, ένα τέλος, μια εισφορά σε ό,τι αφορά τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρωκα. Δύο δις ευρώ θα μπορούσε να μας αποφέρει. Ο φόρος επί της ενέργειας για το διαδίκτυο, για τις, τη τηλεφωνία, το εμπόριο όπλων. Ξέρω ότι οι προτάσεις μου είναι υπερβολικά φιλόδοξες σε σχέση με την ενδιάθεση των ε, κυβερνήσεων. Αλλά η επανευρωποίηση των ευρωπαϊκών πόρων είναι κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Και εκείνοι που πιστεύουν ότι αυτή η πολιτική θίγει την κυριαρχία των κρατών, ε, εγώ θα έλεγα ότι αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης ε, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε κυρίαρχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριο Ντούλιο Ερκολίνο από το Κοινοβούλιο τη Ιταλία. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα τα οποία ήδη ανέφερα κατά την πρώτη συνδιάσκεψη του Οκτωβρίου. Το πρώτο σημείο το οποίο είναι σημαντικό ε, έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπε ο Γάλλος συνάδελφος. Εγώ πιστεύω ότι δεν ε, θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε απέναντι στις αρχές με τι οποίε οικοδομήσαμε την Ευρώπη, να έχουμε περισσότερη Ευρώπη. Γύρω από αυτά, γύρω από αυτή την αρχή θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πιο ρωμαλαίο προϋπολογισμό για την Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχο μου. Ένα πιο ε, ισχυρό προπολογισμό τη Ευρώπη, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερη Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια αρχή ε, απολύτω αδιαφυσβήτητη που θα μα επιτρέψει να ξεπεράσουμε τι αντιφάσει ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέμε και σε αυτά τα οποία πράττουμε όσον αφορά αυτό ε, ε, το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε και που είναι ιστορική σημασία. και εδώ βεβαίω πρέπει να έχουμε ιδίου πόρου. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ε, και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι. Θα ήθελα να σας πω ότι επί τη ουσία συμφωνούμε με αυτά τα οποία ε, ε, ακούσαμε. Θα ήθελα όμως ε, να πω ότι ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, κυρίως όσον αφορά το φόρο επί των κρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ε, για να απαλύνουμε το φόβο ότι δεν θα έχουμε μεταγκαταστάσεις, εκτός δηλαδή μεταφορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της επιβολής του φόρου. Και όσον αφορά το ΦΠΑ, να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε αυτός ο φόρος να μην έχει άνηση επιπτώσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ε, των ε, ε, συντελεστών στα κράτη-μέλη. Στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμα στη διάθεσή μου να σας πω ότι εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους προσωπικούς πόρους αρκεί να έχουμε θάρρος. Πού θα τους βρούμε αυτούς τους πόρους. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την αρχή ενός φόρου που είχε σκεφτεί αρχικά η Επιτροπή ε, όσον αφορά δηλαδή τι εκπομπέ ε, ε, διοξιδίου του άνθρακο. Το φόρο δηλαδή επί των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. Το ανέφερε και ο Γάλλο συνάδελφο. Και η δεύτερη δυνατότητα προέρχεται ανάμεσα στο περιθώριο του μέγιστου των ιδίων πόρων του δημοσιονομικού πλαισίου και των, μη χρησι... των κονδυλίων που δεν χρησιμοποιούνται στον προπολογισμό. Να μην κάνουμε εκεί παζάρια που θα πάρει περισσότερα, που θα πάρει λιγότερα, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά μαζί με άλλα ε, ε, κονδύλια ε, για προϊόντα υψηλή προστέμενη αξία στον τομέα τη έρευνα των υποδομών. δηλαδή, να μην πειράξουμε τι παραδοσιακέ πολιτικέ. Αλλά ποιο είναι το δικό μου το όραμα, ότι με αυτού του συμπληρωματικού πόρου πραγματικά να καταφέρουμε να έχουμε οράματα αριστεία στην Ευρώπη, σχολέ αριστεία, πανεπιστήμια αριστεία, νοσοκομεία αριστεία, τα οποία θα βρίσκονται στην Ευρώπη και θα, και θα δείξουν σε όλου του της Ευρώπης. Τι ακριβώς είναι η Ευρώπη. Γιατί κοιτάξτε, ε, εδώ μιλάμε για τις προοπτικές μέχρι το 2020 και θα πρέπει ε, να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα αυτό ε, χωρίς να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Μπορούμε να τα κάνουμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο περισσότερο θάρρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Τζόργαν Άντερσον, Σουηδία. Από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σουηδική θέση είναι γνωστή. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι όσον αφορά στο δικαίωμα της φορολόγησης. Δεν είναι κάτι που θέλουμε να το αναθέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα παράθυρο, το οποίο είναι λίγο ανοιχτό, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα γιατί φοβόμαστε ότι αυτό θα δημιουργήσει μια κατάσταση την οποία δεν επιθυμούμε. Τώρα για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ακούσαμε ένα επιχείρημα εδώ που λέει ότι από τη μία είναι ένας φόρος και έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις όσον αφορά στις δραστηριότητες που δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους ε, κανόνες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και κάποιοι λένε ότι αυτό είναι κάτι καλό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο αυτό το κεφάλαιο θα παραμείνει εκεί που είναι. Γιατί υπάρχει ένας προφανής κίνδυνος, ενδεχομένως οι δραστηριότητες να είναι διαφορετικές στο μέλλον. Και ο παγκόσμιος αντίκτυπος δεν θα υπάρχει πλέον. Ενδεχομένως να έχουμε στόχους που είναι αντίθετη, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και μια καλή πηγή ισοδύναμος. Ε, εισοδήματος. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με τον ΑΕΠ και η πρόταση δεν είναι αναλογική σε αυτήν την περίπτωση και πρέπει να πω ότι ανησυχώ σε σχέση με αυτό. Αυτό που χρειάζεται τώρα η Ευρώπη είναι περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να επικεντρωθείτε σε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι η πρόταση που έχουμε μπροστά μας εναρμονίζεται με τις αρχές που μόλις ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Merci το λόγο έχει η κυρία Ποδηματά, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρώτη ε, το πρώτο τμήμα της διάσκεψης ε, για τους ίδιους πόρους ε, έχει εξέχουσα σημασία, διότι σχετίζεται άμεσα με το όραμά μας για την Ευρώπη. Και φαίνεται ότι ακόμα και το όραμά μας ε, για την Ευρώπη σε αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης είναι κατακαιρματισμένο. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την άποψή μου, επηρεάζεται υπερβολικά από τις ε, εθνικές ε, χώριες βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες. Ζήτησα το λόγο ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχέδιο γνωμοδότησης για ένα κοινό πλαίσιο ενός ε, φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και η πρώτη διευκρίνηση που θα ήθελα να κάνω εδώ, με αυτή την ευκαιρία, είναι ότι η πρόταση που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος της. Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου προκειμένου να συντονίσουμε διάφορες μορφές και επιλογές φόρων, ε, χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών που υπάρχουν τώρα σε ορισμένα κράτη-μέλη, 9 ή 10. Να συντονίσουμε δηλαδή τις διάφορες μορφές ε, τέτοιων χρηματιστηριακών φόρων, τέτοιων χρηματιστηριακών συναλλαγών αντλώντας μαθήματα από ε, παλιότερα μη επιτυχημένα εγχειρήματα σε αυτόν τον τομέα όπως στην ε, Σουηδία. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι προκειμένου να είμαστε σοβαροί όταν λέμε ότι ε, πάθαμε και πρέπει να μάθουμε, θα πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησαν όλα αυτά. Η χρηματοπιστωτική κρίση που έγινε ε, η οικονομική, νομισματική κρίση. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν ε, να αποφεύγουμε, να μην διορθώνουμε. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι κάλλιστα παρουσίασε όλες τις πτυχές ε, αυτού του θέματος και όπως μπορεί να ξέρετε σε μεγάλο βαθμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, εργαζόμαστε ώστε αυτή η πρόταση να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Ταυτόχρονα, το ξέρω και το ξέρουμε, ότι ότι συνεχίζονται επίπονες συζητήσεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη που ε, έχουν αντίρρηση για την πρόταση, έχουν ε, μεγάλες επιφυλάξεις. Ελπίζω ότι με αυτή τη διάσκεψη θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ε, καλύτερα η μεν τη θέση των δε. Κατά την άποψή μου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να καρποφορήσει αυτή η διάσκεψη. αλλά και γενικότερα όταν ασχολούμαστε με τόσο επιμαχα θέμα όπως είναι ο ε, φόρος για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια για να συζητήσουμε βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και επιχειρημάτων. Και οφείλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε μια λεπτομερέστατη ε, ανάλυση του αντικτύπου που καλύπτει όλες τις ε, πτυχές της εφαρμογής αυτού του φόρου και από την άλλη οι αντιρρήσει και τα επιχειρήματα που ακούγονται εδώ και εκεί. Για παράδειγμα, ότι θα πληγεί η ανάπτυξη, ότι θα έχουμε διαρροή συναλλαγών. Γι' αυτά δεν έχουμε δει μέχρι τώρα απτά συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήματα. Θα βάλω τελεία σε μισό λεπτό. Είναι ένα κύριο θέμα αυτής της συζήτησης ο φόρος για τις συναλλαγές. Ε, ας συζητήσουμε λοιπόν με βάση στοιχεία συγκεκριμένα και επιχειρήματα και ας, αποφύγουμε, ας προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την προπαγάνδα και τα στερεότυπα. Και το τελευταίο τώρα όπως είπε χτες ο πρόεδρος Σούλτς, πραγματικά πιστεύω ότι εμείς οι βουλευτές από τα κράτη-μέλη αλλά και οι ευρωβουλευτές είμαστε σύμμαχοι μεταξύ μας. Και ξέρετε ότι παλιότερα πολλές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόχθησαν για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των αγορών και να αντέξουν την κρίση. Ε, εμείς θα πρέπει να πασχίσουμε για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Και όταν λέμε ότι θέλουμε ο χρηματοπιστωτικός ε, τομέας στην Ευρώπη να υπηρετεί τις κύριες τον κύριο στόχο και την κύρια προτεραιότητα, δηλαδή να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπείς και να τα μεταφράζουμε όλα αυτά σε πραγματικές δράσεις και αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ποδηματά. Το λόγο έχει ο κύριος Κλάστα Άιτχοφ, ε, μέλος ε, του Κοινοβουλίου της, ε, των Κάτω Χωρών. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι Ολλανδός. Καταλαβαίνετε ότι δεν σας εκπλήξει το γεγονός ότι θέλω μετριοπάθεια στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουμε να πληρώσουμε ένα δίκαιο μερίδιο. Το οποίο σημαίνει ότι πληρώνουμε περισσότερα από ό,τι παίρνουμε. Αυτό δεν είναι αποτελεί πρόβλημα από μόνο του. Είναι ένα μερίδιο το οποίο ιδεοδός θα έπρεπε να στηρίζεται απόλυτα στο εθνικό εισόδημα κάθε χώρας μέλους. Εφόσον δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό κατά την άποψή μα σημαίνει σημαντικέ εκτόσει για να εξακολουθεί να είναι δίκαιο. Ε, ε εμένουμε στην αλληλεγγύη ανάμεσα στου Ευρωπαίου, αλλά μην το παρατραβάμε κιόλα. Ε, θα ήθελα να μιλήσω τώρα όχι ω ε, μέλο ε, τη κυβέρνηση τη Ολλανδία και εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ω εκπρόσωπο των πολιτών. Κοιτάξτε, κάθε ευρώ που δαπανάμε, πρώτα απ' όλα προέρχεται από σκληρή δουλειά των Ευρωπαίων. Μην το ξεχνάμε. Και αν πραγματικά θέλετε να αυξηθεί η υποστήριξη για τα καλά που επιφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβετε υπόψη τη βούληση των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτό δεν είναι η δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή που όχι μόνο οι χώρε αντιμετωπίζουν σημαντικέ περικοπέ, αλλά σε κάθε νοικοκυριό οι άνθρωποι υποφέρουν, δεν έχει νόημα να του ζητήσετε να πληρώσουν περισσότερα. Ακόμα και έμεσα, διαμέσου μία σειρά ε, μέτρων που έχουν να κάνουν με νέου πόρου. Ανεξάρτητα από το πώ θα σχεδιάσετε το νέο σύστημα, ε, σε τελευταία ανάλυση ο κάθε Ευρωπαίο πολίτη θα το πληρώσει. Μειώνεται ε, την εθνική συνεισφορά και αυξάνεται την ευρωπαϊκή φορολογία. Αυτό όμω δεν έχει να κάνει με τη μετριοπάθεια που είναι έτοιμα που ζητούν οι πολίτε για τη τελευταία ανάλυση. Πάλι θα τα πληρώσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κώστα Νέβες από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ την ε, Προεδρία και ε, τους συναδέλφους. Και εγώ πέρασα από εδώ και έμεινα και αρκετά χρόνια. Και είμαι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ίδιους πόρους. Πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρει στο να υπάρξει μεγαλύτερη δικαιοσύνη γενικότερα και στην μείωση της της ε, εθνικής συνεισφοράς. Όμως ε, είμαι σκεπτικός έναντι αυτού του ειδικού καθεστώτος που παρέχει το rebate, η έκπτωση. Ε, κοιτάξτε, θα πρέπει να ενισχυθούν, ε, λέμε, τα έσοδα αφενός ε, των ίδιων, από τους ίδιους πόρους. Εδώ βρισκόμαστε σε μία διάσκεψη με εκπροσώπους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο, από το Εθνικά Κοινοβούλιο. Και το θέμα δεν είναι αν θα είναι 5 ή 10% τη εθνική εισφορά. Είναι το 1%. 1% έχει απομείνει. Είναι περίεργο λοιπόν που δεν το βλέπουμε αυτό και δεν μιλάμε για ενίσχυση αυτού του ποσοστού αντί να μιλάμε για μείωση είναι ένα παράδοξο αυτό που γίνεται εδώ. Αφενός λέμε ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την κοινότητα έχουμε περάσει σε ενωσιακό επίπεδο. Όλοι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Θέλουμε σταδιακή ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να διατηρήσουμε τον ίδιο, εάν όχι και ε, μικρότερο προϋπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη στιγμή που μιλάμε για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Για, τη στιγμή, ε, που μιλάμε για περισσότερες θέσεις απασχόλησης και για περισσότερες επενδύσεις. Στην ίδια την ε, πρόταση της Κομισιόν μειώνεται η πρικοδότηση. Ε, είναι αντιφατική αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω ακριβώς ε, πώς έχουν γίνει οι υπολογισμοί εδώ. <clears throat> Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει υπολογιστεί. Μία από τις κύριες προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι η ενίσχυση του προϋπολογισμού, η ενίσχυση των ίδιων πόρων στην Ευρώπη. Μόνο έτσι θα αποκτήσει η Ευρώπη την αξιοπιστία που της αξίζει. Ευχαριστώ. Κυρία Κορνέλια Μιχάλκεν, Αυστρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε εδώ να μπορέσω να μιλήσω σε αυτή την Ολομέλεια. Θα ήθελα να απευθυνθώ, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο από την Ολλανδία που είπε ότι οι πολίτες είναι αυτοί που θα πρέπει, είναι αυτοί που φροντίζουν στην ουσία να πληρώνονται οι ίδιοι πόροι της Ευρώπης, γιατί αυτοί είναι οι φορολογούμενοι και εμείς όλοι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτούς τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά έχω μεγάλες ελπίδες ότι οι ιδέες που θα αναφέρουμε σήμερα ότι θα ληφθούν σοβαρά από τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί έχω λίγο την εντύπωση μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σούλτς, ότι γενικά οι απόψεις είναι ήδη αποκρισταλωμένες. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να εισακωστούμε σε κάποιο βαθμό. Είμαι από μια περιοχή της Αυστρίας όπου η εξοικονόμηση δεν είναι ξένη λέξη, δεν είναι κάτι άγνωστο. Αλλά μπορούμε επίσης να, να, να, προσθέσουμε και άλλες προσεγγίσεις σε αυτή την ιδέα. Γενικά η εξοικονόμηση είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στην Αυστρία. Την επόμενη εβδομάδα οι αυστριακοί πολίτες ε, πρέπει να περιμένουν μεγάλες περικοπές και πρέπει να τις δεκτούν κιόλας και μπορούν να περιμένουν και ότι και η ποιότητα των εξόδων θα πρέπει να ελεγχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά πόσο έχουν νόημα αυτές οι δαπάνες, πού μπορεί να υπάρξει περισσότερη εξοικονόμηση, ποια, είναι τα πραγματικά καθήκοντα στην Ευρώπη, ποια, μπορεί να, ποια προβλήματα μπορούν να επιληθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, πώς διαμορφώνεται πολιτικά η Ευρώπη και πόσο θα κοστίσει αυτό. Άσχετα από αυτό, η Αυστρία συμφωνεί με την πρώτη επιτροπή για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και, και προτιμά μια πιο γρήγορη παρά πιο αργότερα εφαρμογή. Όσον αφορά στο άλλο ζήτημα, δεν βλέπουμε μια προστιθέμενη αξία και δεν θα το υποστηρίζαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόρτας, ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Πορτογαλία, έχετε το λόγο. Στη χώρα μου υπάρχει ένα γνωμικό που αναφέρει κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ε, αυτή η πρόταση δημιουργίας αυτού του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών φτάνει στην Ευρώπη ε, και στους θεσμούς της Ευρώπης, θα έλεγα, με δεκαετίες καθυστέρησης. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, σήμερα ε, έστω και καθυστερημένα, είναι σημαντικό να προσέξουμε ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό. Το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα της πρότασης που παρουσίασε η Επιτροπή είναι ότι ε, με τον τρόπο αυτό ε, θα, θα φορολογηθούν οι συναλλαγές μιας ευρείας γκάμας προϊόντων. Και αυτό είναι το πρώτο θετικό σημείο. Θα ήθελα όμως επίσης, να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ε, περισσότερο κριτική φύσεως. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι ε, το, ε, αυτό το μοντέλο που προτείνεται αφήνει εκτός φορολογίας όλους τους τίτλους ε, που δεν είναι Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκοί, παρόλο που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, ε, διεθνικής επίπεδο Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούμε όσον αφορά την πτυχή αυτή. Δεύτερον, ε, μία άλλη πτυχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο φόρος αυτός θα πρέπει να χρησιμεύσει έτσι ώστε ε, να ε, προωθήσει τα πιο απλά προϊόντα, αν θέλετε, και να τιμωρήσει κατά κάποιο τρόπο τα δομημένα προϊόντα, τα πιο περίπλοκα προϊόντα. Δηλαδή, με δύο λόγια, να φορολογηθούν περισσότερο οι πιο κορδοσκοπικέ συναλλαγέ. Και όμω η πρόταση τη επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στους στόχους αυτούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πρόταση όσον αφορά το σημείο αυτό δεν επιτρέπει να επιληθεί το πρόβλημα της καταπολέμησης της κερδοσκοπίας. Τρίτον, θα ήθελα να ε, απευθυνθώ σε όλους όσους υποστηρίζουν ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα έχει ως συνέπεια διαφυγή εκτός Ευρώπης. Να σας πω ότι το City του Λονδίνου, που είναι το πιο σημαντικό χρηματιστήριο, εφαρμόζει ένα φόρο που είναι σε αυτού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όμως δεν είδαμε διαφύγη κεφαλαίων από το City του Λονδίνου. Και φτάνω τώρα σε αυτό το οποίο με απασχολεί περισσότερο από όλα. Αυτό ο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να χρησιμεύσει ε, για να αυξηθεί η επενδυτική ικανότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Όμως, όπως προβλέπετε τώρα, έχει ως στόχο τη μείωση των εθνικών συνεισφορών στον προπολογισμό. Άρα, λοιπόν, δεν θα επιτρέψει να αυξηθεί η ικανότητα της Ευρώπης να χρηματοδοτεί πολιτικές που δημιουργούν απασχόληση. Θα συμβάλλει στο να μειώσει ε, την εθνική συνεισφορά ε, και ε, τελειώνω εκφράζοντας την επιθυμία να έκανα λάθος και να μην ισχύουν αυτά τα οποία είπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης από την Κύπρο, έχετε το λόγο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί η ε, φορολογία και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα πιο ε, δίκαιο, πιο αποτελεσματικό ένα σύστημα που θα είναι επίσης και αποτελεσματικό. Το νυν σύστημα δεν είναι ε, αποδοτικό αλλά είναι αποτελεσματικό και λειτουργεί. Εάν θέλετε από αυτό το σύστημα να περάσουμε σε ένα άλλο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ σημαντικές πτυχές. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες μικρές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, σίγουρα έχουν πολλά μειονεκτήματα να υποστούν εναντί των μεγαλύτερων και σε αυτές τις χώρες έχουν επινοηθεί ε, φορολογικά συστήματα προκειμένου να αντισταθμιστούν αυτά τα εγγενή, αν θέλετε, μειονεκτήματα που έχουν και να μπορέσουν ε, να επιβιώσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εάν ε, επιβάλλουμε φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μπορεί να σκοτώσουμε τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα σε αυτές τις χώρες και μπορεί να έχουμε πολύ αρνητικό λοιπόν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την οικονομία αυτών των χωρών. Δεν διαφωνούμε με την εφαρμογή ενός φόρου συναλλαγών. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί με μεγάλη προσοχή αλλά και σταδιακά. Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικονομία δεν θα πρέπει να είναι ρηξικέλευτη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά, βαθμιαία. Δεύτερον, μπορούμε να σκεφτούμε διάφορες μορφές φορολόγησης για την χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όπως και ο συνάδελφος ε, από τη Γαλλία, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα είδη φόρων. Εάν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε το ευρωπαϊκό φορολογικό ε, σύστημα, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πολύ προσεκτικά και σε βάθος χρόνου και θα πρέπει να μην εστιαστούμε μόνο σε ένα είδος φόρων. Και ας μην ξεχνάμε και το θέμα των μικρών χωρών. Διαφορετικά μπορεί ε, να οδηγήσουμε σε οικονομική καταστροφή αυτές τις ε, χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούπελ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα την πρόταση του κυρίου Λεβαντόφσκι να τη χαιρετήσω ιδιαίτερα. Νομίζω ότι μας πάει ένα μεγάλο βήμα μπροστά και θέλω να αναφέρω κάποια επιχειρήματα. Πρώτον, είναι μια πρόταση η οποία είναι πιστή στις συνθήκες. Σε όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες η εισαγωγή, η ύπαρξη των ίδιων πόρων ζητείται και προωθείται. Άρα ανταποκρίνεται λοιπόν σε αυτό που αναγράφει στις συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή τίποτα ενάντια στις συνθήκες που έχουμε ήδη συνάψει, ίσα ίσα παραμένουμε πιστοί. Δεύτερον, δεν στρέφεται ενάντια στις αρμοδιότητες των κρατών μελών ή των εθνικών κοινοβουλίων. Όχι, το αντίθετο βασίζεται σε αυτό, στο ότι τα εθνικά κοινοβούλια και το Συμβούλιο ε, οικειοποιούνται αυτή την πρόταση και την υλοποιούν. Και μετά εξαιρετικά θετικό είναι υπέρ του, της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Άλλες αγορές και άλλες επιχειρήσεις τις φορολογούμε, γιατί είμαστε της άποψης ότι μια καλή ρύθμιση των αγορών είναι μια σημαντική συνεισφόρα για την, ε, για την πολιτική. Και υπάρχει τώρα το επιχείρημα, άμα εισάγουμε αυτό το φόρο θα μπορούσε να στραφεί ενάντια της ανταγωνιστικότητας. Εγώ ρωτώ όμως, δεν τον έχουμε. Δεν θα έπρεπε τότε η ανταγωνιστικότητά μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Για μένα ίσα ίσα το αντίθετο θα προκύψει ότι θα πρέπει και τις τράπεζες να τις κάνουμε να συμμετέχουν σε αυτό το ζήτημα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Και είναι ένα κίνητρο για τα κράτη-μέλη να εισπράξουν αυτό το φόρο, γιατί και τα κράτη-μέλη με το ένα θα έχουν ένα τρίτο επιπρόσθετα έσοδα και θα πρέπει να πληρώσουν ε, από μόνα τους κατά 50% λιγότερο. Είναι μια περίπτωση όπου όλοι κερδίζουν και, κερδίζουν και έχουμε και ένα επιπρόσθετο αποτέλεσμα, δηλαδή τα κοινά μας ε, συμφέροντα δεν γίνονται απλώς πολιτική λιτότητας, αλλά προωθούν την ανάπτυξη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά θετική πρόταση και γι' αυτό την υποστηρίζω και όλας πλήρως. Ευχαριστώ. και το λόγο έχει ο κύριος Μίλαν Μάρτιν Σουίκελ, μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου για μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου για τους ίδιους πόρου. Ο κύριος Φίγκελ έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκπρόσωπε ε, του, του Τρίου Προεδρίας, κύριε Λβαντόφσκι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, Μάλιστα το ελεκτικό συνέδριο συμμετέχοντας σε αυτή τη συζήτηση βεβαίως και θα πρέπει να τοποθετηθεί ε, και θεσμικά αλλά και ως ενδιαφερόμενοι. Εμείς πάντως πρέπει να εκδώσουμε γνωμοδότηση ε, για την πρόταση ε, της Επιτροπής. Προετοιμάσαμε την έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες και στην ισοσελίδα μας την προσεχή εβδομάδα και επιτρέψτε μου να σας δώσω ορισμένες, να σας κάνω ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά την πρόταση. Τέσσερι είναι οι βασικέ παρατηρήσει του Ελεκτικού Συνεδρίου για την πρόταση αυτή. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά του νέου ιδίου σπόρου και την πρόταση για, το, για τη βάση του ΦΠΑ συγκεκριμένα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το Ελεκτικό Συνέδριο επέκρινε το υφιστάμενο σύστημα ω ιδιαίτερα πορύπλοκο. Ε, όσον αφορά λοιπόν την κατάργηση του σημερινού συστήματο και από αυτή τη σκοπιά, θεωρούμε ότι το νέο σύστημα θα αντιμετωπίσει τι αδυναμίε του παρελθόντο. Δεύτερον, όσον αφορά το νέο φόρο για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Το συνέδριο σημειώνει ότι η εισαγωγή του φόρου αυτού θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερου πόρου ε, ε, στου εθνικού προπολογισμού, άρα να συμβάλλει στην δημοσιονομική εξυγίανση. Θα συμβάλλει στην δημοσιονομική εξυγίανση. Η πρόταση μεριδίου του φόρου αυτού ω ε, ίδιου πόρου σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί την πρόταση να εφαρμόσουν τον, τον, το φόρο αυτό όλα τα κράτη-μέλη. Εμεί δεν είμαστε αρμόδιοι για να σχολιάσουμε την πιθανότητα ενό τέτοιου εγχειρήματο. Πάντως το νέο σύστημα ε, με, ε, το, το, σύστημα με το, με το εθνικό καφέ προϊόν μέχρι το 2013 ήταν προβλέψιμο. Όμω, ένα νέο ίδιο πόρο ε, από τον καινούριο φόρο θα ε, έχει μια στενή βάση. Γιατί πραγματικά οι, συναλλαγές οι συναλλαγέ αυτέ είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητε. Άρα λοιπόν και ο ίδιο πόρο θα διακυμαίνεται ιδιαίτερα. Τρίτον, όσον αφορά τι εκτόσει ε, και το ζήτημα αυτό, έκτος των εκτόσεων κτλ. Οι ανησυχίε ε, του συνεδρίου αντιμετωπίζονται μέρη στι νέε αυτέ προτάσει. Ε, η καταποκοπή διόρθωση είναι απλούστερη, αλλά εξακολουθεί να μην χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Σημειώνουμε την έλλειψη κριτηρίων όσον αφορά τον προσδιορισμό υπερβολικού δημοσιονομικού άχθου και τέλο, όσον αφορά το κόστο συγκέντρωση των ιδίων πόρων, σημειώνουμε ότι η πρόταση για τη μείωση του κόστου από 25% σε 10% δηλαδή ε, εις βάρος των κρατών μελών. Δεν είναι σαφές το κατά πόσο το ποσοστό αυτό έχει καμία πραγματική σχέση με το πραγματικό κόστος, πάντως θα μπορούσε να προταθεί, να εξεταστεί ε, το κατά πόσο υψηλότερο ε, τέτοιο κόστος θα μπορούσε να, να οδηγήσει, να θαρρύνει τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εκ των υστέρων αξιολόγηση του συστήματος αυτού. Ευχαριστώ. Thank you very much. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Σταβίτσιος ε, είναι αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας για συμμετοχή σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι όλες οι ιδέες που ακούγονται σήμερα και όλες οι απόψεις που εκφράζονται εξ ονόματος εθνικών κοινοβουλίων θα εισακουστούν από εκείνους που χαράσουν πολιτική και ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν άμεσα. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι συνθήκες όχι μόνο στο σκέλος έσοδα αλλά και στο σκέλος έξοδα, δαπάνες του προπολογισμού. Αυτή είναι μια οικουμενική αρχή ε, που ακούμε συνεχώς και εδώ και θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή αυτής της αρχής. Η ευρωπαϊκή απόφαση για, την, ε, για τους νέους πόρους, ίδιους πόρους, είναι πολύ σημαντική και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητά μας πια, θα πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σωστά και να κάνουμε και μία μελέτη αντικτύπου ε, για αυτή την απόφαση. Ο φόρος ΦΠΑ τώρα φτάνει γύρω στο 11%. Όμως το διοικητικό κόστος για την ίσπραξη είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα έσοδα από αυτόν τον πόρο. Οι επιβαρύνσεις λοιπόν μετά το 2014 σε αυτό το επίπεδο το διοικητικό θα πρέπει να μειωθούν. Ε, Επίση, ε, δεν είναι πλήρω εναρμονισμένος ε, ο φόρος ΦΠΑ. Ε, λόγω τη κρίσης, κάποιοι αύξησαν τον ειδικό αυτό φόρο. Η βάση είναι διαφορετική μεταξύ κρατών μελών. Θα θέλαμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για να προωθηθεί η εναρμόνιση. Και περιμένουμε βεβαίως και μία μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα επηρεάσουν όλα αυτά τους καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις, δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ε, διορθώσεις. Θα μειωθούν πώς, κατά το ίμιση, ελπίζουμε. Ελπίζουμε, έχουμε πολλές ε, και μεγάλες φιλοδοξίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να επιμείνουμε. Τέλος, δεν πιστεύω ότι οι νέοι φόροι θα σώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σωθεί με μια αποτελεσματική ε, και χρηστή διαχείριση. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Ευχαριστώ. Κυρία Μουλμπάχα από την Αυστρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ την πρόταση της Επιτροπής τη βλέπω ως μια βάση διαπραγμάτευσης. Αλλά εδώ να μην ξεχάσουμε σε, σε ποια πλαίσια βρίσκονται τα, τα μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση έχει στοιχήσει πάρα πολύ στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Και εμείς ε, στην Αυστρία έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά μέσα του προϋπολογισμού για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και για να αναζωογονήσουμε την οικονομία. Και, με αυτό το πλαίσιο, και σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω την εισαγωγή, τουλάχιστον την πρόταση εισαγωγής ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών οι χρηματοπιστωτικές αγορές και στην Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρουν. Όχι μόνο οι μεμονωμένες σε οικονομίες και μεμονωμένα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ, γιατί πολλές φορές τα κέρδη ε, ήταν ιδιωτικοποιημένα, αλλά τα χρέη δημόσια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ να υπάρξει συνεργασία όλων των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βλέπω μια σοβαρή εξέλιξη σύμφωνα με την οποία η πολιτική δεν ε, δείχνει αυτή την πρόθεση διαμόρφωσης ε, που θα ήθελε. Δεν μπορεί να διαμορφώσει την πολιτική έτσι όπως θέλει. Αλλά η πολιτική εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Και γι' αυτό, αγαπητές κυρίες και κύριοι, απευθύνω την έκκληση, αυτή την, αυτό τον φόρο πραγματικά να το συζητήσουμε καλά, να δούμε όλα τα υπέρ, όλα τα κατά, να τα ζυγίσουμε όλα. και να συζητήσουμε ξανά αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι στην Ευρώπη περιμένουν από εμά τους πολιτικούς, περιμένουν λύσεις. Λύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και λύσεις όσον αφορά την κοινωνική ευζοία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη, την απασχόληση των νέων, ε, διάφορα ζητήματα. Κλείνοντας, επειδή έχει αναφερθεί πολλές φορές αυτό το σχόλιο, για το μηχανισμό διόρθωσης. Η Αυστρία πλήττεται από μια αλλαγή αυτού του μηχανισμού διόρθωσης. Πάρα πολύ σύντομα η Αυστρία μπορεί να φανταστεί μια τέτοια αλλαγή με καταποκοπήν ποσά αν για όλα, αν είναι ισότιμη η μεταχείριση όλων των κρατών. Και αυτή τη στιγμή η πρόταση δεν βαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες από το ΕΛΚ, το Κοινοβούλιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, ε, να σας χαιρετήσω όλους και να σας συγχαρώ για την διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης όπου συμμετέχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό ε, είναι κάτι που ενδιαφέρει και τα δύο μέρη. Ε, και για, για παράδειγμα όσον αφορά την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού ε, και εκεί πιστεύω ότι αν είχαν εμπλακεί ε, και, και τα εθνικά κοινοβούλια, το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό και τον προπολογισμό, ε, να πω το εξή. Πιστεύω ότι ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσουμε και να καταλάβουμε τη λειτουργία του προπολογισμού σε σχέση πάντα με τις εθνικές συνεισφορές. Μιλήσαμε για απλότητα, απλούστευση, για διαφάνεια. Είναι πήγον να ακολουθήσουμε την οδό αυτή για να μπορέσουμε και όλοι να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Εδώ συμφωνούμε όλοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, όλοι θέλουμε το σύστημα να είναι πιο απλό και να τεθεί τέρμα σε αυτό το σύστημα ε, επιστροφών, ε, επιστροφής που, με το οποίο διαφωνούμε. Όσον αφορά τώρα την πρόταση του ίδιου πόρου τη Επιτροπή, ναι, αλλά ε, εδώ πρέπει να το δούμε το θέμα σε συνδυασμό με, την, με περισσότερη αλληλεγγύη που απαιτείται. Πρέπει λοιπόν να, τεθεί, να δοθεί ένα τέλο στη διάκριση ανάμεσα στους καθαρούς δικαιούχους και στους καθαρούς συνεισφέροντες. Πραγματικά και το θέμα της δίκαιης επιστροφής, αυτό το «gist retour» που λέτε στα γαλλικά, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει. Δεδομένη της κατάστασης των εθνικών προϋπολογισμών, ε, σήμερα ε, μιλάμε για πλαφόν 1%. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω μία ευχή σύντομα να πάμε στο 1,23% ε, του ε, ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για να ενισχύσουμε τελικά αυτόν τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτός, ε, μην ξεχνάμε, ότι είναι επενδύσει, ο επενδυτικός προϋπολογισμός, Το μεγαλύτερο του μέρος αφορά επενδύσεις. όταν λοιπόν μιλάμε για επενδύσεις, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, τότε σίγουρα θα πρέπει να καταλήξουμε στο λογικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό. Μα νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχο ε, και του συστήματο των ιδίων πόρων. Μιλήσαμε πολύ για ανάπτυξη σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Μιλήσαμε πολύ για επενδύσει. Ε, ε, ε, είμαι διπλά ικανοποιημένο, αλλά μην ξεχνάμε την οικονομική συνοχή, την εδαφική συνοχή, την κοινωνική συνοχή. Όλα αυτά δεν θα μπορέσουν ποτέ να γίνουν στι πλάτε και ει βάρο τη συνοχή. Όσον αφορά τώρα αυτόν τον ε, φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρε που διστάζουν ιδιαίτερα. Εδώ επιτρέψτε μου να θέσω το εξή ερώτημα. Απέναντι στην ε, αδυναμία που υπάρχει να συμφωνήσουν όλοι με την ιδέα αυτή. Ε, ποια είναι η εναλλακτική λύση, τι θα γίνει δηλαδή αν δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα ερώτημα προς την Επιτροπή. Ο κύριο Σανκάουερ από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την ε, συζήτηση. Θα θυμάστε όλοι σας ότι ήταν δύσκολο να υιοθετηθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Η εφαρμογή της όμως εστεύθη με επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να ακολουθήσουμε το άρθρο 311 που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της. Ε, σε περίοδο βέβαια οικονομικής ε, κρίσης ε, και δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά. Έχουμε εδώ μία πρόταση ε, σωστή, νομίζω, για ε, τους δύο νέους ίδιους πόρους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σαφές, εύληπτο και διαφανές σύστημα για τους πολίτες μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιες ε, ερωτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν για ε, τον φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών σίγουρα θα πρέπει να εξεταστούν οι συνέπειές του στην ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών εάν υπάρξει διαρροή τέτοιων συναλλαγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ε, κανόνας θα ισχύσει της εγκατάστασης ή της συναλλαγής ε, και ποια θα είναι η επιβάρυνση για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Λάσσε Μπράντετ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πράσινους. Κυρία Μπράντεν, συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά μου σωστά. Ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που έχουν έρθει από τις πρωτεύουσές τους σήμερα, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη συζήτηση από κοινού. Και τώρα, για αυτόν τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, κατά την άποψή μα, είναι απλώ μια άλλη μορφή ΦΠΑ. Γιατί πιστεύουμε ότι αν αγοράζει έναν καφέ ή αγοράσει ε, ένα αυτοκίνητο και πληρώνει φόρου, πληρώνει φόρου για όλε τι συναλλαγέ. Ο μοναδικό τομέα που δεν πρέπει να πληρώσει φόρου όταν υπάρχει συναλλαγή είναι ο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και δεν βλέπουμε τώρα τη διαφορά γιατί ένα τομέα πρέπει να φορολογείται και ένα άλλο όχι. Και υπό αυτή την έννοια, για για μας είναι ένας από τους λόγους ύπαρξης αυτού. Και τώρα το ερώτημα, θα ποινικοποιήσει μια χώρα ή μια πόλη περισσότερο από την άλλη. Νομίζω ότι η πρόταση που έκανε η Επιτροπή είναι πάρα πολύ έξυπνη. Και δεν ανοίγει την πόρτα για κάτι τέτοιο, αλλά βρήκε έναν τρόπο και νομίζω μετά από πάρα πολύ μελέτη και σκέψη και προσπάθεια να αποφύγει ακριβώς αυτή την παγίδα και να το κάνει πολύ πιο ελκυστικό για όλους τους συμμετέχοντες. Και μετά, πού πάνε τα χρήματα. Μέχρι τώρα η πρόταση λέει το 1 τρίτο πάει στον εθνικό Προϋπολογισμό άμεσα και τα 2 τρίτα πάνε στον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό μειώνοντας κατά 50% τις Εθνικές Συνεισφορές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό 100% επιστρέφει στα κράτη-μέλη στην ουσία. Και μετά, αυτό που είπε ο Ολλανδός συνάδελφος, κάνει καμία διαφορά αυτό για τους πολίτες μας τι πληρώνουν και πού. Ναι, έχει μια διαφορά γιατί φορολογούμε φορολογούμε ένα τομέα που δεν έχει φορολογηθεί μέχρι τώρα και νομίζω ότι αυτό θα επιτρέψει μια καλύτερη δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο χωρίς να βελτιώσει την ε, δυνατότητα ε, επένδυση στην, ε, στην ανάπτυξη, στην αλληλεγγύη στο ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να μειώσουμε το χρέο μα και να συνεχίσουμε να μπορούμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη με το να συνεισφέρουν όλοι αυτοί που είναι μέρο του οικονομικού συστήματο. Και γι' αυτό το λόγο ότι πραγματικά θα ήταν καλό αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό από κοινού. Ενδεχομένως να υπάρξουν ακόμα κάποιες αλλαγές, αλλά νομίζω είναι ένας καλός τρόπος ε, διαφυγής και νομίζω ότι θα αποφελήσει τους πολίτες μας σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Πριν ξαναδώσουμε το λόγο στους, στα μέλη του πάνελ, η κυρία Ισαμπέλ Τουιρόν, αντιπρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλο τη Ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είμαι τελευταία παίρνω το λόγο, επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία έτσι ώστε να απευθυνθώ ω μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στα μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου. Ε, σε εσά που εκπροσωπείτε τα εθνικά κοινοβούλια, τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Οι στιγμέ που ζούμε σήμερα είναι ιδιαίτερε Δεν είναι η πρώτη φορά που, που συναντιόμαστε βεβαίω και συνεργαζόμαστε, αλλά είναι αρκετά σπάνιο θα έλεγα ε, κάτι τέτοιο. Και επευθύνω έκκληση έτσι ώστε στα κοινοβούλια σα, ε, στους διαδρόμους των κυβερνήσεων που προετοιμάζουν δύσκολους προπολογισμού και αυτό γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη, να μπορέσετε να εξετάσετε αυτή την καλή πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι Όλοι μαζί, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, καλή πρόταση τη Επιτροπή, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό που μα προτείνεται σήμερα, το ακούσαμε πολλέ φορέ, είναι και σωστό, αλλά και αποδοτικό και αποτελεσματικό. Σας παρακαλώ λοιπόν να εξετάσετε αυτή την πρόταση με ρεαλιστικό πνεύμα ε, προ το συμφέρον και των εθνικών μα προπολογισμών, γιατί και εγώ ε, προέρχομαι από μια χώρα που πρέπει να ληφθούν δύσκολα μέτρα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύτιμη ευκαιρία να κάνουν περισσότερα, καλύτερα και κυρίω να τα κάνουμε μαζί. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν στι επιτροπέ σα, ε, στα εθνικά σα κοινοβούλια, στην Επιτροπή Προπολογισμού, στην Επιτροπή Οικονομικών να εξετάσετε με ρεαλιστικό πνεύμα ε, πέραν ιδεολογικών σκέψεων την πρόταση αυτή, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και του εθνικού προπολογισμού και τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που με τι επενδύσει του ε, θα ξαναγυρίσει στα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν εμεί οι Ευρωπαίοι και εσεί ε, που προέρχεστε από τα Εθνικά Κοινοβούλια να δράξουμε την ευκαιρία. Για πρώτη φορά τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε μια καλή πρόταση. Είναι ιστορική σημασία στη στιγμή και θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με με, ε, τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά πειθαρχήσατε και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, πρώτα απ' όλα στον κύριο Λεβαντόφσκι, τον Επίτροπο, που φαντάζομαι ότι έχει πολλά να πει μετά από όλες τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Αυτά όλα αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε τέτοιες ε, συναντήσεις. Πρέπει να επικοινωνούν οι αιρετοί ε, από όλα τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Να σας πω το εξής. Ε, ακούσαμε μεγάλο βαθμό υποστήριξης προς τις προτάσεις της Επιτροπής και νομίζω από την πλειοψηφία των ομιλητών. Αλλά ε, επιτρέψτε μου να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε αυτές ε, τις επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, ερωτήσεις που αναφέρθηκαν. Ξεκινώ από τα δύο μέλη ε, του πάνελ, τον κύριο Μαυρογιάννη και την κυρία Χάνσεν που, ε, ε, Αντρέα, έχουμε δύσκολες συζητήσεις για τον προπολογισμό. Επίσης, ε, ε, ε, θα ήθελα να αναφερθώ και στους δύο συναδέλφους από τη Σουηδία και από τις κάτω χώρες. Δύο χώρες που επί τη ευκαιρία ε, είναι χώρες που θα δοθούν διορθώσεις. Και βεβαίως δεν μπορούμε να εγκινηθούμε σαφώς καθαρή θέση όσον αφορά τις ροές και τις εκροές με βάση τις δαπάνες. Δεν μπορούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε ε, μία δίκαιη θέση μόνο διαμέσου των δαπανών που να αντικατοπτρίζει και τον πλούτο των χωρών αυτών. Άρα απαιτούνται κάποιες διορθώσεις. Εξού και η πρόταση για τις αιτήσει διορθώσεις, που αυτή η πρόταση, ε, οι διορθώσεις ε, είναι αναγκαίες για τις δύο αυτές χώρες, αλλά και για το Ευρωπαϊκό, και για, την, και για το Ηνωμένο Βασίλειο, που, όπου προβλέπεται και έκπτωση, αλλά και για τη Γερμανία. ο κύριο, η κυρία και ο κύριο Πόρτα, ο κύριο Μαυρίδης, ο κύριο Σοκάουερ εξέφρασαν κάποιε επιφυλάξει, ε, ε, ε, ερωτήσεις και να ήθελα να σας πω και να, το εξή και να επαναλάβω ορισμένε βασικές ιδέες. Η πρότασή μας για τους ιδίους πόρους ε, παρακολουθεί ιδιαίτερα και το πνεύμα και το γράμμα των Πιστεύουμε στην δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών. Ε, καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση. Αυτό αποτελεί και την ε, ε, βασική μου θέση. Αυτό που θέλουμε είναι να θέσουμε επιτάπητος την πρόταση και μετά από τις συζητήσεις τα εθνικά κοινοβούλια θα αποφασίσουν. ενώ πρέπει να υπάρξει ομόφωνη κύρωση οποιασδήποτε πρόταση για φορολογία. Η πρότασή μα για του ε, ίδιου πόρου δεν έχει ω στόχο την αύξηση του προπολογισμού. Η πρότασή μα για το χρονικό διάστημα 2014-2020 είναι μετριοπαθή και πρέπει να πω ότι ακούσαμε και κριτικέ για το γεγονό ότι είμαστε μόλι το 1%. 1,18% ήταν στη δεκαετία του 1990. Ε, τώρα, η πρότασή μας για τις πληρωμές για το επόμενο διάστημα στηρίζεται στο 1% παρά, το, παρά τη συμφωνία μας ε, στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Δηλαδή, είπαμε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη εν ώψη του ορίζοντα 2020. Ε, Εξετάσαμε λοιπόν, όπω σα είπα, το μακροσκελή κατάλογο υποψηφιωτήτων για του ίδιου πόρου και προσπαθούσαμε να δούμε τι είναι πιο αποδοτικό, τι είναι πιο δίκαιο και τι αποτελεί πραγματικά νέο εισόδημα. Και εδώ είχαμε την κυρία Μπράτνερ ε, για ένα, που εξέφρασε απόψη για ένα τομέα που δεν είχε φορολογηθεί. Διότι δεν προβλεπόταν ε, για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, κανένας φόρος. Ενώ η Ευρώπη πρέπει να πούμε ότι ε, συμβάλλει ιδιαίτερα για τη διατήρηση ενό υγιού χρηματοπιστωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το κριτήριο ακολουθήσαμε για την επιλογή του συγκεκριμένου πόρου. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εθνικέ πρωτοβουλίε. Όπω σα είπα, 10 χώρε ήδη φορολογούν ε, τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Και θα ακολουθήσουν και άλλε, αυτό είναι σίγουρο. Ε, ακούσαμε και αυτό το οποίο είπε η κυρία Ποδηματά. Ε, το θέμα. Δεν είναι ε, κατά πόσα θα φορολογήσουμε αυτές τις συναλλαγές. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Ε, εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καλό για να αντιμετωπίσουμε και τις ανταγωνιστικές τρευλώσεις. Καλύτερο να έχουμε μια εναρμονισμένη βάση. Έτσι ώστε να μειωθούν και οι εθνικέ συνεισφορέ, γιατί εδώ μιλάμε για προσπάθειε που καταβάλλονται σε όλε τι χώρε για εξυγίανση των προπολογισμών. Και όλα αυτά γίνονται με βάση την εμπειρία μα. Δεν είμαστε ε, αφελείς. Ε, ε, παρακολουθούμε και το τι έγινε στη Σουηδία. Να σα πω ότι εμένα μου αρέσουν οι πρωτοβουλίε που παίρνει η χώρα αυτή σε πολλού τομεί. αλλά ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν εύκολο το σύστημα που ακολουθήθηκε αυτή τη φορά. Ε, υπήρχε μεγάλη δυνατότητα ε, ε διαφυγής. Ε, δηλαδή, επειδή είχε ως βάση τον τοπικό ενδιάμεσο, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε κανείς να αλλάξει με γραφείο, να πάει στο εξωτερικό και να διαφύγει, να, φορο, να υπάρξει φοροδιαφυγή. Μελετήσαμε λοιπόν ιδιαίτερα τι έγινε στη Σουηδία η ίσπραξη του φόρου ε, θα γίνεται ε, με βάση ε, την έδρα και την εγγραφή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μέρος πηγαίνει στον εθνικό προϋπολογισμό, άρα όσο περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχουν στη χώρα, αυτό το 1 τρίτο θα είναι μεγαλύτερο το 1 τρίτο του φόρου. Και τα 2 τρίτα θα, ε, ε, θα προορίζονται για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αλλά και εδώ θα μειωθούν οι εισφορές με βάση την κλίδα ε, ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Γι' αυτό μιλήσαμε για 50% μείωση. Ε, η μείωση θα γίνει αυτόματα με βάση το, ε, το κλειδί, ε, την κλίδα ακαθάριστο εθνικό προϊόν και όχι με βάση αυτά που εισπράττονται στα κράτη-μέλη. είναι τεχνικό το ζήτημα, ιδιαίτερα δεν πρόκειται να επισέλθω σε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Αλλά να σα πω τώρα, ήθελα να τα πω όλα αυτά με βάση τον αντίκτυπο. Τώρα, εμείς μιλάμε ε, για ε, αυτόματες ε, ε, βραχυπρόθεσμες συναλλαγές που γίνονται με βάση, ε, τους, ε, ε, με βάση ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και πρέπει να, να δούμε ότι εδώ είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε τον αντίκτυπο όταν έχουμε να κάνουμε με αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση. Πρέπει να δούμε όμως το πώς η αρχή της έδρας και της εγκατάστασης ε, θα μειώσει ε, τον κίνδυνο διαφυγής. Και πιστεύω ότι τώρα η αξιολόγηση αντικτύπου χαρακτηρίζεται από περισσότερη ισορροπία. Η πρώτη ήταν μονόπλευρη. Είχε να κάνει με το τι θα μπορούσε να συμβεί και πάλι στην πραγματική οικονομία βεβαίω. Τι θα μπορούσε να συμβεί με την εισαγωγή αυτής, της, αυτού του χρηματοπιστωτικού φόρου. Αλλά αν μιλάμε για 81 δις, γιατί αυτές είναι οι προβλέψεις μας, ε, 81 δις από το φόρο αυτό, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της φορολογίας σε άλλους τομείς και να ε, ανακουφίσουμε τη φορολογία της εργασίας. Άρα η, ε, ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία ε, ξεκινά με ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο. Και Γι' αυτό έχουμε αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου, για το γεγονό ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Είναι, ε, κατά την άποψή μου, είναι η μέθοδο που θα οδηγήσει στην μικρότερη ζημιά στην πραγματική οικονομία. Επίση, έγιναν πολλές παρατηρήσεις ε, για τον εμετάβλητο χαρακτήρα. Είπε και το ελεκτικό συνέδριο ε, κάποια πράγματα. Εδώ όμω έχουμε και το αντιστάθμιμα με τις εθνικές συνεισφορέ. για την αντιστάθμιση αυτού που είναι περισσότερο ευμετάβλητο και πώς να το πω, ε, λιγότερο σταθερό. Όταν μιλάμε για τελωνιακούς δασμούς, ε, ίδιους πόρους, φορολογία, πάντα έχουμε τον παράγοντα μετριασμού, τον παράγοντα αντιστάθμισης που είναι ακριβώς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Όσον αφορά τις διορθώσεις, δεν πρόκειται να επισέλθω στο ζήτημα αυτό ιδιαίτερα, οπότε δεν μου απομένει παρά να σας ευχαριστήσω όλους ε, ε, για την τόσο πλούσια και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Θα τα λάβουμε όλα αυτά που είπατε υπόψη και ε, ελπίζουμε να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά και εμείς θα βελτιώσουμε την πρότασή μας με βάση τη δική σας συνεισφορά. Ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για όλες τις απόψεις που ακούσαμε σήμερα. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε αυτές τις συνεισφορές ή ε, να ξέρουμε ποιες είναι οι άλλες απόψεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και είναι σαφές ότι δίστανται οι απόψεις για αυτά τα θέματα. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον ε, Άντερς που είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνουμε τέτοιου είδους διαλόγους. Είναι πολύ σημαντικό να συναντιόμαστε και να επιδιώκουμε στο μέλλον περισσότερες συναντήσεις τέτοιου είδους όπως είπε και εσύ, η είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Ευρωβουλευτών και Εθνικών Βουλευτών. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρατήρηση. Και η κυρία μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Βέλγιο μας είπε να πάμε πίσω στα εθνικά μας κοινοβούλια και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση κυρίως ε, επί της προτάσεως που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί είναι και δίκαιη και αποτελεσματική αυτή η πρόταση. Εδώ όμως νομίζω ότι συνεχίζουμε να έχουμε κάποια προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ στη δική μου παρουσίαση προσπάθησα να ε, πιέσω τον Επίτροπο να μας πει περισσότερα πράγματα για τον αντίκτυπο αυτών των προτάσεων. Θα πρέπει να, να μάθουμε ε, περισσότερα πράγματα για τις συνέπειες αλλά και για τον καταμερισμό των βαρών. Εντάξει, μιλάμε για την αλληλεγγύη, μιλάμε για το ποιο θα πρέπει να πληρώσει, αλλά δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε. Το ξέρω από τι συζητήσει που κάνουμε και σε εθνικό επίπεδο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ε, τις ίδιες ε, πληροφορίες και την ίδια τεκμηρίωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να κάνουμε συνείδητα αυτή τη συζήτηση ε, και σε εθνικό επίπεδο. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτή την έκκληση είναι ο μόνος τρόπος αυτός για να έχουμε μία βάση για μία εντελεχή συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια. Και έτσι μπορείτε, ε, μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς περισσότερο. Και αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρώπη σήμερα. Θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Θα πρέπει να γνωρίζουν περισσότερο τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ευχαριστήσω και την Αν Γένσεν για την εισαγωγή της. Χαίρομαι διότι συμφωνούμε επί των αρχών και αυτό είναι πολύ καλό. Ε, ανήκουμε και στην ίδια πολιτική παράταξη. Δεν είμαστε ε, μόνο ε, από την ίδια χώρα. Και εγώ λοιπόν όπως και εκείνη θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να δούμε περισσότερο την ποιότητα των δαπανών αυτή τη στιγμή, σήμερα στον προϋπολογισμό. Ο Ολλανδός συνάδελφος είπε ότι μιλάει εξ ονόματος των πολιτών. Ως ερετή ε, βουλευτές όλοι μιλάμε εξ ε, των ε, πολιτών και ιδιαίτερα των ψηφοφόρων μας. Αλλά αυτόν τον διάλογο θα πρέπει να τον κάνουμε ανοιχτά και να είμαστε διαφανείς για την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξουν αυτά τα έσοδα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στο τι κερδίζουμε, στην προσθέμενη αξία. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες μας. Ποια είναι τα αποτελέσματα από τους διάφορους τίτλους του προϋπολογισμού και Πού χρειάζονται αλλαγές. Νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό λίγο περισσότερο και ελπίζω ότι όλα θα διευκρινιστούν λίγο περισσότερο και στην απογευματινή συζήτηση. Γιατί και αυτή ε, μας αφορά στη συνέχιση των συζητήσεών μας για τους ίδιους πόρους. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Κυρία Τζένσεν, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η αξία μιας τέτοιας συζήτησης είναι ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει το πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην παρερμηνεύουμε ο ένας τον άλλον. Και είναι σημαντικό για μένα να είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητά τους ίδιους πόρους προκειμένου να αυξήσει τις δαπάνες, αλλά ζητά τους ίδιους πόρους προκειμένου να υπάρξει ένα πιο διαφανές σύστημα για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβετε ότι εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση και γνωρίζουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη και που θα αντιμετωπίσουν και για πολλά χρόνια ακόμα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής κρίσης. Γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα των δαπανών. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα δεν είναι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οροφές επί του προπολογισμού. Στην ουσία περιορίζουμε το, ε, τον ετήσιο, τους ετήσιους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο μέχρι το 2020. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε και ενδεχομένω να αναρωτηθείτε κατά πόσο τα όρια που θέλατε να βάλετε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ανταποκρίνονται στα όρια που θα βάζατε στον εθνικό προϋπολογισμό κατά πόσο θέλετε να εισαγάγετε κάτι παρόμοιο όπως και αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Ευρώπη, η Επιτροπή περιορίστηκε στα ποσά που παρουσίασε. Είναι στην ουσία ένα απαράλλαχτο όριο από το 2013 έως το 2020. Είναι μεγάλος περιορισμός σε έναν ε, προϋπολογισμό ο οποίος ε, ενδέχεται να εμπεριέχει νέα καθήκοντα, διευρύνσεις, νέα πράγματα που θα γίνουν. Και όλοι λέμε ότι χρειάζεται να βρούμε αρνητικές προτεραιότητες, αλλά έχω ανακαλύψει ότι από τη στιγμή που κάποιος πρέπει να βρει αρνητικές προτεραιότητες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Ιδιαίτερα γιατί πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Και νομίζω ότι η Επιτροπή προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο στην πρότασή της και να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα. Ένα μεγάλο μέρος συζήτηση σήμερα έγινε για το φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όταν, συζητήσαμε αυτές τις, όταν αρχίσαμε τις συζητήσεις αυτές το 2008-2009, πολύ σοβαρά στο Κοινοβούλιο, νομίζω ήταν μια πλειοψηφία κατά. Και αυτό σταδιακά έχει αλλάξει. Τώρα έχουμε μια πλειοψηφία υπέρ. Και είμαι στην περίεργη κατάσταση εγώ να είμαι μέρος της μειοψηφίας ενάντια στο φόρο αυτό. Αλλά ακόμα ακούω τον Γιάννος και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που προσπαθεί να μου εξηγήσει. Αλλά σίγουρα θα υπερασπιστώ το ότι χρειαζόμαστε νέους ίδιους πόρους. Ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι μια επιλογή. Υπάρχει βέβαια και το ΦΠΑ και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια έντονη συζήτηση επί αυτού του θέματος αλλά κατά την, κατά την άποψή μου είναι ένας ισχυρός υποψήφιος για ίδιους πόρους που εμπεριέχει και μια ε, απλούστευση, απλοποίηση του συστήματος και ενδεχομένως και καλύτερο έλεγχο του ΦΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν σε σχέση με την πρόταση για το ΦΠΑ και ακόμα δεν έχουμε, συζητήσει, δεν έχουμε αρχίσει αυτή τη συζήτηση. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ε, ε, δούμε. Από τη Γαλλική Γερουσία αναφέρθηκε ότι υπάρχουν ενδεχομένω και άλλες ε, πιθανότητες. Ναι, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε και αυτή τη συζήτηση. Ακούσαμε ε, για την ενέργεια, αλλά μπορώ να φανταστώ και άλλες επιλογές όπου μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή και για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε αυθεντικούς ίδιους σπόρους για την Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον συζητώντας αυτά τα ζητήματα. Το δύσκολο πράγμα φυσικά είναι ότι αυτό πρέπει να αποφασιστεί μεταξύ των κρατών μελών με ομοφωνία. Δεν είναι μια εύκολη συζήτηση, αλλά θα πρέπει να δούμε τα κράτη-μέλη να ακούν το ένα το άλλο και να κλείνουν το ένα προς το άλλο. Σίγουρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να διευκολύνουμε αυτή τη συζήτηση με το να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματα όπως το κάναμε και σήμερα και να βοηθήσουμε και τη συζήτηση και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ επικοδομητικό. Κάτι τελευταίο. Μετά με ενέπνευση η Αυστριακή συνάδελφος που θα λέγοντας ότι θα μπορούσαμε να πάμε κάποια πράγματα πίσω στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε ωστόσο να εξοικονομήσουμε και δαπάνες για τα εθνικά κοινοβούλια κάνοντας κάποια πράγματα από κοινού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε στα εθνικά κοινοβούλια. Ενδεχομένως να μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση με το να γίνουν από κοινού κάποια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε μια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ασχολείται με τις αερογραμμές, την ασφάλεια των αεροπορικών ταξιδιών. Υπάρχει μία ε, υπηρεσία που πιστοποιεί τα αεροπλάνα και τα πληρώματα. Εκεί που παλιά είχαμε 27 τέτοιες υπηρεσίες. Σίγουρα πρέπει να υπήρξε κάποια εξοικονόμηση από αυτό. Δεν ξέρω αν τα Εθνικά Κοινοβούλια βρήκαν αυτές τις εξοικονομήσεις. Σε κάθε περίπτωση γυρίσεις πατρίδες σας και βρείτε. Βρείτε τις. Ας πούμε, οι συζητήσει για την υπηρεσία εξωτερική δράσης. Ξέρω ότι στη δική μου χώρα η υπηρεσία αυτή έχει προκαλέσει μια συζήτηση στη Δανία για το πόσο πραγματικά χρειάζεται να επενδυθεί στις, ε, στα, στις πρεσβείες εφόσον υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρεσβεία. Και πράγματι εδώ βρίσκουμε εξοικονόμηση εξαιτία τη κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να δούμε μόνο τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω μια δαπάνη, αλλά μπορεί επίση να είναι και ένα μηχανισμό εξοικονόμηση δαπανών για τα εθνικά κοινοβούλια και τα και τους εθνικούς προϋπολογισμούς και, και προτείνω να γυρίσετε στις πατρίδες σας και να το σκεφτείτε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρογιάννης εξ ονόματος Συμβουλίου έχει το λόγο. Ε, Πολύ σύντομα και εγώ πιστεύω ότι ε, έχει ξεκινήσει τώρα η συζήτηση, ε, έχει ξεκινήσει με τα καλά, για τα καλά θα έλεγα. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί με ανοιχτό πνεύμα και να λάβουμε υπόψη βεβαίως τη σημερινή πραγματικότητα, τις σημερινές πραγματικότητες. Εργαζόμενοι με μια βάση και μια προσέγγιση γνήσια ρεαλιστική. Όπως είπε η κυρία Γιάντσεν, σήμερα η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στο φόρο πρέπει ενδεχομένω ε, να μην αρκεστούμε σε αυτό, αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε ανοιχτό πνεύμα, όπω άλλωστε υπογράμμισαν πολλοί από του ε, ε, συναδέλφου που πήραν το λόγο, και θα πρέπει να μην αποκλείουμε εκ των προτέρων τίποτα. Να εξετάσουμε και άλλε δυνατότητε. Και σήμερα έγιναν πολύ ενδιαφέρουσε υποδείξει. Πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο εάν σεβαστούμε προφανώς τις αρχές της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης και όσον αφορά τους πόρους ε, και τις δαπάνες, τα έσοδα δηλαδή και τις δαπάνες και δεν λέω ότι υποστηρίζω την αρχή της γνήσιας επιστροφής, όχι. Αν αυτό καταλάβατε, ε, δεν θέλω να τοποθετηθώ ούτε για το ούτε στο συγκεκριμένο σημείο αυτό δεν θέλω να αναφερθώ. Ε, Πάντω ε, πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να μην κάνω τώρα σχόλια επί τη ουσία όσον αφορά τι επιμέρου θέσει ε, όπω αναπτύχθηκαν. Σίγουρα εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, αλλά πιστεύω ότι στους προσεχείς μήνες όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και σε εθνικό επίπεδο κυρίως να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση με τα νέα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν σήμερα, ενδεχομένως να ε, κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια ε, και επεξήγησης σε εθνικό επίπεδο. Και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν βάσιμε ελπίδες ε, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πριν το τέλος του χρόνου και να φτάσουμε σε μια λύση που θα είναι ικανοποιητική και σύμφωνοι ε, με τις, ε, και με τις αρχές της συνθήκης αλλά και με τις προσδοκίες ε, των πολιτών μας. Πιστεύω ότι η Ιδανική Προεδρία θα προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο αυτό το δύσκολο θέμα. Εμείς που θα πάρουμε τις σκητάλη στη συνέχεια Ελπίζουμε να μην ε, έχουν μείνει πολλά για να κάνουμε εμείς, όμως βεβαίως και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε ε, τον καλό δρόμο που ε, έχουμε διανύσει όλοι μέχρι στιγμής. Δεσμευόμαστε με όλη μας την καρδιά και όλα τα όργανα, όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμευόμαστε έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια λύση που θα είναι στο ύψος των κοινών προσδοκιών μας. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο, ε, να κάνει μια σύντομη ερώτηση ένα σύντομο σχόλιο ε, προς, τα μέλη του πάνελ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πεινάμε όλοι. Πολύ ωραία την κατάλληλη στιγμή, γιατί έχουμε την ευγενική πρόσκληση Δανική Προεδρία σε ένα γεύμα, το οποίο ε, θα γίνει δύο ρόφου πιο κάτω στο ίδιο αυτό κτίριο. Σας παρακαλώ όμως να είστε στην ώρα σας ε, ε, για την απογευματινή συνεδρίαση στις 2.30 ακριβώς. Καλή όρεξη σε όλους.